Muy buenos días. Bonjour à tous. Καλημέρα σας. Good morning. <laughs> Muy buenos días. We should be kicking off. Ας ξεκινήσουμε. Ως συνήθως έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη και πρέπει να ξεκινήσουμε υπενθυμίζοντας πόσο μεγάλη σημασία έχει ο χρόνος. Αρχίζω από τις ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Πρώτα απ' όλα για κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει στην ημερήσια διάταξη. Η πρώτη είναι ότι δεν θα ψηφίσουμε την έκθεση Χολμάγερ για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών. Θα είναι ανταλλαγή απόψεων επί των τροπολογιών και όχι ψηφοφορία. Δεύτερον, η συζήτηση μέλο για την Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας έχει αναβληθεί. Δεν θα είναι εδώ εισηγητή σήμερα γι' αυτό. Τρίτον, η γνωμοδότηση Χάνκης όσον αφορά την προστασία συστημάτων θα συζητηθεί, που δεν συζητήθηκε χτες, θα συζητηθεί σήμερα για την προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας στις 11 και 4. Να έχετε υπόψη σας ότι στις 9 Φεβρουαρίου οι συντονιστές με πλειοψηφία αποφάσισαν να ζητήσουν άδεια για έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας όσον αφορά την κατάσταση στην Ουγγαρία και ζητούν την αντίστοιχη επιτροπή από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ε, κάποιες ομάδες ζήτησαν βάσει του άρθρου 192 του κανονισμού να ζητηθεί έγκριση. Η έγκριση αυτή προβλεπόταν για τις 10 σήμερα το πρωί. Αλλά ξέρετε ότι υπό το φως της έγκρισης που έγινε στην Ολομέλεια της έκθεσης για τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία. Μιλάω για το Στρασβούργο, έτσι, 16 Φεβρουαρίου, εκεί. Πριν από λίγες μέρες δηλαδή, πριν από δύο εβδομάδες. Βάσει λοιπόν αυτής της έγκρισης, πιστεύουμε ότι η έγκριση στην Επιτροπή μας δεν είναι πλέον αναγκαία, εφόσον η Ολομέλεια έχει ήδη αποφασίσει. Συνεπώς, το σημείο αυτό αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη μια που συμφωνούν και οι συντονιστές ότι η έγκριση δηλαδή εδώ στην Επιτροπή μας δεν είναι πλέον αναγκαία εφόσον υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας. Θα υπάρξει ψήφισμα για την ε, κατάσταση στην Ουγγαρία, της πολιτικής εξελίξεις εκεί. Τέλος, να σας υπενθυμίσω ότι κυρία Γκέπαρτ και η γνωμοδότησή σας γνωμοδότησε Κάσμαν όσον αφορά τις συνέπειες ε, ιδιοκτησίες έχει αναβληθεί για την επόμενη συνεδρίασή μας 21η Μαρτίου. Συνεπώς, χωρίς άλλη καθυστέρηση, περνάμε στο σημείο 9, που είναι το πρώτο ουσιαστικό σημείο που έχουμε σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Υπενθυμίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας για κάθε ένα από τα σημεία που θα εξετάσουμε, γιατί συνεδριάζουμε σήμερα το πρωί και το απόγευμα, αλλά στο μεταξύ θα υπάρξει και συνεδρίαση των συντονιστών στις 12.30. Εάν λοιπόν θέλουμε να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη μας για να προλάβουμε να εξετάσουμε όλα τα θέματα στο χρόνο που τους έχει δοθεί. Σημείο 9 λοιπόν όπως έλεγα, σχετικά με την τροποποίηση του κώδικα συνόρων Σέγγεν και τη σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Σέγγεν. Η συγγετής μας είναι ο συνάδελφος Γεώργιος Το σημείο αυτό έχει να κάνει με τη συζήτηση των τροπολογιών που έχουν υποβληθεί από το, στο σχέδιο έκθεσης του κύριου Παπα-Νικολάου. 39 εκθέσεις. Θα ακούσουμε λοιπόν τον εισηγητή μας και μετά θα έχουμε συζήτηση. Πρέπει όμως να σας πω ότι στόχος μας είναι να έχουμε και μια ψηφοφορία προς ανατολισμού 20 και 21 Μαρτίου, ώστε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις για μια πρώτη συμφωνία. Παρακαλώ έχετε το λόγο κύριε Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας. Για να επανέλθουμε στη συζήτηση του θέματος αυτού, το οποίο είναι τεχνικό κατά κύριο λόγο. Οι τροπολογίες τελικά δεν είναι τόσο πολλές. Είχαν υποβληθεί όντως 39 τροπολογίες, κάποιες αυτές από τον ίδιο τον εισηγητή και οι υπόλοιπε από τα διάφορα, τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ τους σκιώδες εισηγητές για τόσο καλή συνεργασία που είχαμε μεταξύ μας για αυτό το θέμα. Την κυρία Μπόσκορ, την κυρία Βέμπερ, την κυρία Ένστε, την κυρία Στάνοκα και τον κύριο Κίρκοπ. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέρφους που επέβαλαν τροπολογίες, τον κύριο Κοέλιο, την κυρία Χολμάιερ και την κυρία Μακοβέη. Επιτρέψτε μου να, συ... να έρθω εδώ στη συζήτηση ενός θέματος που συζητήθηκε και στην προηγούμενη συζήτηση. Είναι το, 21 Δέλτα που μιλάει για τη δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη να αναφέρουν την παρουσία υπηκών τρίτων χωρών στις ε, χώρες τους. Κάποιες χώρες λοιπόν το κάνουν ήδη. Αυτή είναι η τρέχουσα κατάσταση στο κάτω-κάτω της συνθήκης Σέγγεν. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο πρέπει να καταγράφονται στους δήμους τους οι υπήκοοι τρίτων χωρών. Μόνο η Δανία, η Ιταλία, η Λιθουανία και η Εστονία δεν έχουν εφαρμόσει το άρθρο αυτό 22 της ηθίκης του Σέγγεν. Οι άλλες χώρες το έχουν κάνει με διάφορες εθνικές νομοθεσίες τους. Γι' αυτό και αν ακόμα και αν στην αρχή λέγαμε ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό αυτό το μέτρο, η Επιτροπή που παρακολουθεί αυτό το θέμα λέει ότι δεν χρειάζεται διάταξη αυτή γιατί στην πράξη δεν λειτουργεί. Ε, λέει να μην είναι υποχρεωτική. Και εμείς λέμε όντως τα κράτη-μέλη να αποφασίζουν τι θέλουν να κάνουν. Θα ήθελα επίσης εδώ να υπογραμμίσω ότι στην τροπολογία μας 22 επανισάγουμε για άλλη μια φορά την αρχή της ε, αμοιβαιότητας όσον αφορά τα ταξιδιωτικά έγγραφα. Ο κύριος Κοέλιο, ο κύριος Έγκεν όπως τον ονομάζουμε, το είπε αυτό. Η προσέγγιση μας είναι ίδια κατά κάποιο τρόπο με το Συμβούλιο, αλλά σας υπενθυμίζω ότι εδώ έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε μια διαφορετική γραμμή για τους ελέγχους στα σύνορα, για να είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Παρόλο λοιπόν που είχαμε ίδια προσέγγιση αντίστοιχη με το Συμβούλιο, δεν θέλουμε να τα βάζουμε μαζί τις φραγίδες της θεωρήσεις και όλα. Μετά από συζητήσεις πάντως με τον κύριο Κοέλιο, είπαμε ότι θα έπρεπε να ευθυγραμμιστούμε με τις άδειε παραμονής. Είναι σημαντικό λοιπόν να προβλέπετε κάτι τέτοιο εδώ. Τώρα για τις άλλες τροπολογίες. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι τροπολογίες δεν δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα και πιστεύω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε κάποια συμφωνία και σε βιβασμό εξού και οι τροπολογίες οι συμβαστικές. Οι 53, 54 και 56 για τα εξωτικά έγγραφα της κυρίας Μπόσκορτ που μιλάνε για τρίτων χωρών στην πράξη καταλαβαίνουμε γιατί θέλει την τροπολογία αυτή και μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι για να μπορούμε να υπολογίσουμε τη διάρκεια διαμονής του τρίτου υπήκου είναι σημαντικό το τοξιδιωτικό έγγραφο να σφραγίζεται και όταν μπαίνει στη χώρα και όταν βγαίνει από τη χώρα το άτομο αυτό. είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούμε να κάνουμε έναν έγκυρο υπολογισμό. Τώρα, αν δεν έχει σφραγίδα εισόδου το άτομο, τότε μπορούμε να υποθέσουμε ότι παράνομα μπήκε στην επικράτεια του κράτους μέλους. Το ίδιο ισχύει αν λείπει και μια σφραγίδα εξόδου. Πάλι οι αρχές μπορούν να θεωρήσουν ότι ο υπήκος τρίτης χώρας μπήκε τέλος πάντων παραμένει παράνομα στην επικράτεια του κράτους μέλους, οπότε σύμφωνα με την αντίστοιχη οδηγία πρέπει να μπορεί να επιστρέψει στην χώρα προέλευσής του. Και εδώ πολύ θα ήθελα να ακούσω και την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερον, για το θέμα των ε, ε, σημείων από όπου μπαίνουν ε, μετανάστες στις χώρες. Εδώ είναι αναγκαίο η επικράτεια της χώρας όπου βρίσκεται το σημείο αυτό να είναι είτε στο κράτος μέλος είτε σε τρίτη χώρα. Οι συνάδελφοι από την ΚΟΕ λένε ότι ένα τέτοιο σημείο κοινό ε, πρέπει να είναι μόνο σε χώρες μέλη. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω καλύτερα ε, το επιχείρημα, αλλά αυτό που έχω να σχολιάσω είναι η έννοια των ε, διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες, γείτονες τρίτες χώρες, είναι ακριβώς να ελέγχονται τέτοια κοινά σημεία διέλευσης από όπου μπαίνουν ή βγαίνουν μετανάστες, σύμφωνα με την νομοθεσία της άλλης χώρας. Ε, πιστεύουμε, εγώ τουλάχιστον πιστεύω, ότι δεν θα είναι εφικτό εφόσον τέτοια σημεία ε, θεωρούνται μόνο σημεία που βρίσκονται στις χώρες μέλη. Δεν μπορώ να φανταστώ οι χώρες μέλη να μπορούν να συμφωνήσουν στο Συμβούλιο. Επιπλέον, έτσι φτάνω και στην τροπολογία 58 της κυρίας Δανόκα που λέει ότι το, κράτο, το υπήκος μάλλον τρίτης χώρας περνάει παράνομα δεν μπορεί να ελεγχθεί βάσει του παρόντος κανονισμού. Κάποιος ο οποίος έχει ήδη περάσει ή αυτός ο οποίος προσπαθεί ή υπάρχει πόνοια ότι προσπαθεί ή θα προσπαθήσει να περάσει. Εδώ η διάκριση όπως καταλαβαίνετε όπως λεπτή και έχει να κάνει με άτομα τα οποία βρίσκονται στην επικράτεια τρίτου, τρίτης χώρας. Αν πάντως κάποιος βρεθεί παράνομα να περνάει, πρέπει να πάει στον πλησιέστερο σταθμό φύλαξης. Αλλά ποιο είναι αυτός. Είναι εκείνο ο οποίο βρίσκεται στην επικράτεια της χώρα μέλους ή είναι εκείνο ο οποίο βρίσκεται στην επικράτεια της τρίτης χώρα. Και εμείς λέμε ότι πρέπει να βρίσκεται είτε στη χώρα μέλο, είτε στην τρίτη χώρα. προκειμένου να ελεγχθεί και να εντοπιστεί ποιος ακριβώς ε, είναι αυτός που προσπαθεί να περάσει τα σύνορα. Για την εποπτεία τώρα, ξέρω τις θέσεις των συναδέλφων, αλλά είναι σημαντικό εδώ να ξέρουμε ότι εφόσον δεν έχουμε αποτελεσματικά μέτρα εποπτείας και ελέγχου, δεν μπορούμε να έχουμε και έναν αποτελεσματικό χώρο Σέγγεν. Τέλος, υπάρχουν και πολλές τροπολογίες από την ε, ΚΟΕ και τους σοσιαλιστές που έχουν να κάνουν με το σημείο 632 για τους ελέγχους όσον αφορά τους ελέγχους σε λεωφορεία κλπ. Οι συνάδελφοι της ΓΟΕ θέλουν να διαγραφεί η διάταξη αυτή, ενώ οι σοσιαλιστές θέλουν να παραμείνει ως δυνατότητα και όχι ως υποχρέωση. Ε, περιμένουμε ότι θα συζητήσουμε και θα καταλήξουμε σε συμβασμούς για αυτά τα θέματα. Αυτές είναι κάποιες από τις τροπολογίες κλειδί. Από εκεί και πέρα περιμένω τους συναδέρφους να πούνε τι σχόλια έχουν και τι παρατηρήσεις. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε καρποφόρα συζήτηση σήμερα μέχρι την ψηφοφορία, την προσανατολισμού που θα κάνουμε σε κάνα μήνα. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε την τόσο καλή συνεννόηση που είχαμε μέχρι τώρα. Θέλω να ακούσω και τα σχόλια και της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Για άλλη μια φορά, ευχαριστώ ε, όλους και το, την Προεδρία της Δανίας και την Επιτροπή και όλους όσοι συνεργάστηκαν τόσο καλά μαζί μου για αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ακούμε τους εκπροσώπους της Επιτροπής και του συμβουλίου Είναι εδώ και θέλουν να λάβουν το λόγο. Παρακαλώ. Η Επιτροπή έχει εκπρόσωπο. Παρακαλώ, είστε εδώ. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήδη στην προηγούμενη μας συνεδρίαση είχαμε υπογραμμίσει ότι η συντριπτική πλειονότητα των τροπολογιών που έχει καταθέσει ο κύριος ε, Παπα-Νικολάου μας φαίνονται ικανοποιητικές και μπορούμε να τις δεχτούμε ίσως πλην τη 42. Τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στη 43 με 81, τις λοιπές τροπολογίες δηλαδή. Και τις ε, προτάσεις που έχουν να κάνουν με την ε, διεξαγωγή ελέγχων σε πλοία, είτε σε εγχώρια ύδατα, είτε στην ανοιχτή θάλασσα προτάσεις οι οποίες βλέπουμε ότι δεν απαιτούνται. Επισημάναμε λοιπόν ότι στην έκθεση του κυρίου Παπα-Νικολάου και στις νέες τροπολογίες ορισμένες δεν μας γεννούν δυσκολίες τους προς την ουσία. Ωστόσο βλέπουμε ότι ξεπερνούν το πεδίο εφαρμογής αυτής της τεχνικής μάλλον προσαρμογής και γι' αυτό θα θέλαμε να περιοριστούμε στα ζητήματα που έχουμε να εξετάσουμε εδώ για να προχωρήσουμε γρήγορα σε ένα καλό αποτέλεσμα. Οι τροπολογίες αυτές, Φερρυπίν, είναι η 59, η οποία αναφέρεται στις συνέπειες της άρνησης εισόδου, που είναι ενδιαφέρουσα, αλλά δεν ανήκει στο πεδίο εφαρμογής της προτάσεως άλλες τροπολογίες. Θα είχαν θέση μάλλον στο πλαίσιο της πρότασης για τη διακυβέρνηση Schengen και όχι σε αυτή την νομοτεχνικής φύσεως προσαρμογή για τον κώδικα. Η παραδείγματι η τροπολογία για τον ορισμό της απειλής για την εσωτερική ασφάλεια που είναι ενδιαφέρουσα πρόταση αλλά πάλι δεν έχει θέση τεχνο... τεχνικού χαρακτήρα αυτή προσαρμογή. Άλλες τροπολογίες ξεπερνούν το πεδίο του κώδικα συνόρων Σέγγεν, Φερρυπίν, η υπαριθμών 63 έως και 66 οι οποίες προτείνουν την διεύρυνση των εγκληματικών ε, δραστηριοτήτων υπό την έννοια της Συμφωνίας Σέγγεν, δηλαδή δεν σχετίζονται με τον κώδικα, για δε τα τις 67 με 72 τροπολογίες που έχουν να κάνουν με την ε, με τα κοινά σημεία διάβασης, κοινά συνοριακά σημεία διάβασης. Πιστεύουμε ότι είναι ενδιαφέρουσε. θα πρέπει να προσπαθήσουμε σε συνεργασία με τους συντάκτε τους να ε, δούμε λύσεις, γιατί έχουν ενδιαφέροντα στοιχεία και μπορούμε να καταλήξουμε σε συνενετικές λύσεις. Και όπως είπα, στα κοινά αυτά σημεία διάβαση των συνόρων είναι απαραίτητο να έχουμε καλούς, σαφείς κανόνες. Η Επιτροπή θα πρέπει λοιπόν να επαληθεύσει τις θημερείς ε, συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών και τρίτων κρατών για αυτά τα κοινά σημεία ελέγχου. Αλλά για να το πράξει αυτό χρειάζονται σαφεί κανόνε και σαφεί κατευθυντήρε γραμμέ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι απαραίτητο αυτό. Και επίση, όπω όπως ήδη επεσήμανε ο κύριο Παπα-Νικολάου, ορισμένε από τι νέε ε, τροπολογίε, 53 57 παραδείγματι και 76 έως 89 ε, σφράγιση και προϋποθέσεις, μάλλον προδιαγραφές ε, στα θαλάσσια σύνορα. Αυτή τη στιγμή διαπιστώνουμε ότι αντίκυνται στον κώδικα, στο βασικό πνεύμα του κώδικα και γι' αυτό θα τις απορρίπτουμε διότι μπορεί να υπονομεύσουν ολόκληρο το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ κύριε Λούτς. Και τώρα το Συμβούλιο παρακαλώ αν θέλει να λάβει το λόγο. Είστε εδώ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ και καλημέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον εισηγητή αλλά και τους σκιώδεις ε, εισηγητέ της Επιτροπής σας ε, που προέτειναν ε, τροπολογίες. Η Προεδρία θεωρεί ότι αποτελεί καλή βάση για διαπραγματεύση και το σχέδιο έκθεσης και οι τροπολογίες. Ε, η συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι δυνατή και πριν από το τέλος της Προεδρίας μας. Και τι, η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου δεν είχε ακόμη την ευκαιρία να εξετάσει διεξοδικά το σχέδιο εκθέσεως και τις τροπολογίες. Η γενικότερη αίσθηση που επικρατήσει επί του Συμβουλίου Αντίστοιχα μετά όσα είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι πως οι τροπολογίες στο σχέδιο κανονισμού δεν θα πρέπει να ξεπερνούν το πεδίο που καλύπτει η αρχική πρόταση της Επιτροπής. Όσον αφορά το Συμβούλιο, απαραίτητο είναι να επιτευχθεί εν ευθέτω χρόνο συμφωνία προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή σύντομα νέες διατάξεις που θα διευκολύνουν συνθήκες για τους ε, συνοριοφύλακες, θα εξασφαλίζουν ένα σαφές πλαίσιο για τους ταξιδιώτες και θα ορίζουν σαφείς ε, διαδικασίες. Η διαδικασία λοιπόν τώρα στο Συμβούλιο δείχνει προς μια γενική συμφωνία ότι η τροποποίηση του άρθρου 5 παράγραφος 1 θα πρέπει να ε, ισχύσει για τους ε, ταξιδιώτες χωρίς προξενική θεώρηση αλλά και για τους υπηκόους τρίτων κρατών για τους οποίους απαιτείται θεώρηση διαβατηρίων. Και έτσι λοιπόν αντίστοιχα θα πρέπει να τροποποιεί το άρθρο 5 σε παραπομπή, σε σχετισμό μάλλον με τον κώδικα ε, θεώρηση διαβατήριων. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παπα-Νικολάου και τα μέλη της Επιτροπής σας για την πολύ καλή συνεργασία. Τέλος, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε στους προσεχείς μήνες μια καλή συμφωνία στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος, και τώρα συζήτηση. Έχουμε ένα σχετικά βραχή κατάλογο ομιλητών. Ο κύριος Κοέλιο έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστώ τον κύριο Παπα-Νικολάου, ο οποίος έκανε μια πολύ καλή έκθεση. Και έτσι ξεκίνησε τα λόγια του ε, επισημένοντας ότι πρόκειται για μια τεχνικού χαρακτήρα έκθεση. Ε, δεν ε, παρέλειψε να κάνει και πολιτικές τοποθετήσεις γιατί οτιδήποτε έχει να κάνει με τα σύνορά μας έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, είναι ευαίσθητο θέμα και ως εκ τούτου πολιτικό θέμα. Τον ευχαριστώ θερμά για την πολύ καλή συνεργασία και τη συνοχή τη έκθεση αυτή με προηγούμενε τοποθετήσει του Κοινοβουλίου μας, όπως σε παραδείγματι θεώρηση μακρά διαρκεία, προξενική θεώρηση μακρά διαρκεία και άλλα αντίστοιχα ζητήματα. Εν είναι καλή η έκθεση, είδα τροπολογίες που κατέθεσε ο ίδιος ο κ. παπα την βελτιώνουν, βελτιώνουν ακόμη περισσότερο την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ελσιού. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, μιλήσω εκ μέρους του σκιώδου μας, ο οποίος δεν ε, μπορεί να είναι εδώ σήμερα δυστυχώς. Ευχαριστούμε τον κύριο Παπα-Νικολάου ήταν πολύ καλή η συνεργασία, πολύ καλός ο συντονισμός του έργου στην έκθεση αυτή. Και θα ήθελα να επισημάνω ότι στόχος των τροπολογιών που καταθέσει η δική μας ομάδα ήταν η προστασία, η διαφύλαξη της ελευθερίας κυκλοφορίας των πολιτών μας μέσα στο χώρο Σέγγεν. Και γι' αυτό δεν συμφωνούμε και δεν θα συμφωνήσουμε ούτε και θα υπερψηφίσουμε η αδίποτε τροπολογία ή που θα οδηγεί σε περιορισμό ή περιστολή αυτών των θεμελιωδών ελευθεριών. Μέσα σε αυτή την έκθεση. Η, έκθεση, η ομάδα μας υποστηρίζει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο μας από την έκθεση αυτή την κατάρτιση σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα για τους συνοριοφύλακες. Η κατάρτιση αυτή πρέπει να περάσει, πρέπει να εγκριθεί. Οι σύνοριοφύλακες δηλαδή θα πρέπει στο μέλλον να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ευχερός ποια είναι τα ευάλωτα άτομα που χρήζουν βοηθείας. Για δε τα κοινά σημεία ε, ελέγχου στα σύνορα θέλουμε να επανέλθει η αρχική πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβανομένης υπόψη ιδιαίτερα όμως της ανάγκη για προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και παρακαλούμε τον εισηγητή να διευκρινίσει την θέση του ως προς τις τροπολογίες που δεν έχουν άμεσο συσχετισμό με την ε, έκθεση αυτή που είναι τεχνικού χαρακτήρα, επί παραδείγματος της υπαριθμών 63, 64 και λοιπές τροπολογίες. Θα ήθελα να τοποθετηθεί όπως αυτό ο εισηγητής μας. Μια τελική παρατήρηση. Έλεγχη σε πλοία, νιοψίες, ανάλογα με, την, ε, με τη διάσταση του κινδύνου για την ασφάλεια, τη λαθρομετανάστευση, θα πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Thank you very much. Η κυρία Βέμπερ, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομη. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω αυτά τα οποία είχα πει στην πρώτη συνομιλία μας. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς τον κύριο Παπα-Νικολάου για τον τρόπο με τον οποίο έκανε δεκτές τις θέσεις μας στα πλαίσια της προετοιμασίας και κατάθεσης της πρότασής του. Αυτά τα οποία μένει να γίνουν από εδώ και πέρα είναι κυρίως να προσπαθήσουμε να δούμε εάν υπάρχει δυνατότητα να υπάρξουν συμβιβασμοί σε ορισμένες από τις τροπολογίες και ταυτόχρονα να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε από κοινού το τι δεν είναι δεκτό στην έκθεση αυτή γιατί ξεπερνάει την εμβέλεια της έκθεσης και γι' αυτό η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι χρήσιμη. Νομίζω ότι τα πλαίσια του ιδίου πνεύματος συνεργασίας που επεδείχθη μέχρι τώρα ε, θα υπάρξει περαιτέρω επικοινωνία με τους κοιόδης και τους εισηγητές. Η κυρία Στάνοκα. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ, λέει η κυρία Στάνοκα, τον κύριο Παπα-Νικολάου για τον τρόπο με τον οποίο οργάνωσε τη διαδικασία αυτή και τον τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκε με τους σκιώδεις εισηγητές και κατέθεσε την πρότασή του. Φυσικά εμείς υποστηρίζουμε τις προτάσεις τις οποίες κάνει σχετικά με τις τεχνικές λεγόμενες τροπολογίες. Υπάρχουν κάποια θέματα προς συζήτηση ακόμα γιατί δεν συμφωνούμε με το υποχρεωτικό της αναφοράς, η κοινοποίηση και ζητάμε την κατάργηση αυτής της πρότασης, αυτή είναι η δική μας θέση. Σχετικά με τη δική μας τοπολογία την 58. Ο κύριος Παπα-Νικολάου εξέφρασε τις αμφιβολίες του σχετικά με τον μηχανισμό που προτείνεται για την εφαρμογή αυτής της πρότασης. Κοιτάξτε, αν μπορούμε να βρούμε μια καλύτερη διατύπωση, γιατί όχι. Αλλά αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς βασίζεται ουσιαστικά σε κάποιες προτάσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν για να δοθούν νομικές εγγυήσει σε αυτούς οι οποίοι ζητούν διεθνή προστασία. Ίσως θα ήταν βέβαια δυνατό να αποφύγουμε κάποιες παρανοήσεις και να προσπαθήσουμε να προτείνουμε διακόπτη η ομιλήτρια να προτείνουμε ένα ορισμό ο οποίος να μην ερμηνεύεται με διαφορετικό τρόπο κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Εν πάση περιπτώσει το θέμα αυτό θέλει δουλειά ακόμα και θα προσπαθήσουμε. Πάντως θέλω να ευχηθώ στον κύριο Παπα-Νικολάου να συνεχίσει να είναι αποτελεσματικός και παραγωγικός. Η κυρία Μάκινταερ. Τελευταία ομιλήτρια και μετά θα δώσω το λόγο στον εισηγητή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παπα-Νικολάου για τη δουλειά που έκανε μέχρι τώρα. Η πολιτική μου ομάδα έχει δύο πεδία ανησυχίας. Το πρώτο αφορά το θέμα ασφαλείας αξιολογούμε θετικά τη συμπερίληψη της τροπολογίας 36 που λέγει ότι η πρόσβαση στα συστήματα πληροφόρησης ε, από τρίτες χώρες και από εκπροσώπους τρίτων χωρών θα απαγορεύεται. Αυτό είναι θετικό και το εκτιμούμε ιδιαίτερα. Ο άλλος τομέας που μας απασχολεί είναι η αύξηση του κόστους και του γραφειοκρατικού βάρους, αν θέλετε, στα κράτη-μέλη. Σαν παράδειγμα αυτό το οποίο προτείνεται στην τροπολογία 17 λέγεται ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να δίδονται σε μια γλώσσα η οποία να γίνει επαρκώς κατανοητή από το πρόσωπο το οποίο ε, υφίσταται τη διαδικασία. Έτσι και αλλιώς έχουμε πει ότι οι πληροφορίες θα πρέπει να δίδονται σε κάθε γλώσσα της Ένωσης και της τρίτης χώρας, στα σύνορα της οποίας ε, υπάρχει το συμβάν. Οπότε θα πρέπει να προσπαθήσουμε εδώ να μην αυξήσουμε χωρίς κάποιο ε, επαρκή λόγο το διοικητικό βάρος. Κύριε Παπα-Νικολάου έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Είναι τιμή μου που καταλήγουμε νομίζω σε μια συμφωνία. Οι αποστάσεις ανάμεσα στις διαφορετικές θέσεις που εκφράστηκαν δεν είναι τόσο μεγάλες Σχετικά τώρα με τα σχόλια τα οποία ακούστηκαν, προφανώς θα υπάρξει τις επόμενες μέρες μια συνάντηση των σκιωδών. Προφανώς θα έρθουμε σε επαφή με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για περαιτέρω συζητήσεις. Τώρα να απαντήσω σε κάποια θέματα τα οποία ίσως ε, ε, να ξεπερνούν αν θέλετε την έκθεση αυτή. Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας εμείς ακολουθήσαμε τη συγκεκριμένη γραμμή από την αρχή. Από την αρχή είπαμε ότι δεν θέλουμε να ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας. Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τα πάντα. Θέλουμε να παραμείνουμε σε ένα τεχνικό επίπεδο, ταυτόχρονα όμως να συμπεριλάβουμε και κάποιες πολιτικές παρατηρήσεις και ευχαριστώ εδώ τον κύριο Κοέλιο για αυτά που είπε, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο λειτουργίας του SBC, του Schengen και της Σύμβασης γενικότερα. Νομίζω ότι καταφέρνουμε να διατηρήσουμε μια κάποια ισορροπία. Η απόκρισή μας λοιπόν είναι σαφής. Δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε την εμβέλεια της συγκεκριμένης έκθεσης. Ακόμα και αν κάποια από τα σχόλια που ακούστηκαν είναι ενδιαφέροντα, Ίσως θα πρέπει να συμπεριληφθούν σε κάποια άλλη έκθεση, σε κάποιο άλλο έγγραφο, σε κάποια άλλη συζήτηση, όχι σε αυτήν εδώ. Συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Λούτς για τους ξεκάθαρους κανόνες που θα πρέπει να υπάρχουν στα πλαίσια της λειτουργίας του SBC. Είναι σαφές ότι δεν πρέπει να συγχαίουμε, να δημιουργούμε συγχύσεις στα κράτη-μέλη και θα ήθελα να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις ε, με το Συμβούλιο σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης. Νομίζω ότι έχουμε μια σταθερή βάση διαπραγμάτευσης πλέον και αυτά θα τα δούμε λεπτομερέστερα τις επόμενες εβδομάδες. Έχω κρατήσει κάποιες ε, παρατηρήσεις εδώ. Ξέρω δεν έχουμε πολύ χρόνο για να δώσω πλήρεις απαντήσεις να πω ότι σε σχέση με τους ε, συνοριοφύλακες και την εκπαίδευσή τους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήδη έχουμε καταθέσει αντίστοιχες τροπολογίες, είναι πολύ σημαντικές οι τροπολογίες αυτές. Κανένας ε, δεν μπορεί να αρνηθεί ότι η Σέγγεν σημαίνει ελεύθερη διακίνηση στα πλαίσια του Σέγγεν. Πρέπει να προστατεύσουμε την αρχή αυτή και δεν πρέπει να επιτρέψουμε διαφορετικές ερμηνείες που θα δημιουργήσουν συγχύσεις και δεν θα ξεκαθαρίσουν το μήνυμα. Ευχαριστώ και την κυρία Βέμπερ για τα σχόλιά της και για το πνεύμα συνεργασίας που εξέφρασε από την αρχή. Την ευχαριστώ που δεν κατέθεσε τροπολογίες. Την ευχαριστώ για την ειλικρίνειά της είχε συγκεκριμένα σχόλια. Τα σχόλια αυτά συμπεριελήφθησαν στην πρώτη πρόταση και την ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ εν πάση περιπτώσει όλους τους συναδέλφους. Θα παραμείνουμε σε στενή επαφή τις επόμενες εβδομάδες. Θα έχουμε πολλές συναντήσεις για να κλείσει επιτέλους το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Είμαστε στο χρόνο που προεβλέπετο, λέει ο Πρόεδρος. Ένα τελικό θέμα είναι ότι θα πρέπει λοιπόν να συζητήσετε τις τροπολογίες, τις συναντήσεις σας με τους κοιόδης εισηγητές, έτσι ώστε να προχωρήσουμε σε μια ψηφοφορία προς ανατολιστικού τύπου στις 21 Μαρτίου για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Περνάμε στο επόμενο θέμα το οποίο είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα σχετικό με ε, την διαδικασία Schengen. Είναι ο κανονισμός 562 του 2006 για τη θέσμηση κοινών κανόνων με την προσωρινή επαναφορά ελέγχου στα εσωτερικά σύνορα σε εξωτερικές περιπτώσεις. Η συγγήτρια είναι η συνάδελφος Ρενάτε Βέμπερ, η οποία θα πάρει το λόγο για να ξεκινήσει η συζήτηση. Μετά θα ακούσουμε τις απόψεις των άλλων οργάνων, Προεδρία και Επιτροπή και θα, γίνει, θα μείνει και χρόνος για συζήτηση. η επόμενη, η συζήτηση μπορεί να κρατήσει την επόμενη ώρα. Η κυρία Βέμπερ έχει το λόγο. Καταρχάς θα ήθελα να εξηγήσω στους συναδέλφους και να ζητήσω συγγνώμη μάλλον από τους συναδέλφους γιατί προς το παρόν η έκθεση αυτή υπάρχει μόνο στα αγγλικά μου. Ε, με είχαν διαβεβαιώσει ότι μέσα σε αυτή τη βδομάδα θα είχαμε όλες τις γλώσσες. Ελπίζω λοιπόν στο τέλος της εβδομάδας να έχετε τη δυνατότητα πριν καταφέσετε τροπολογίες να εξετάσετε την έκθεση αυτή στη μητρική σας γλώσσα. Αυτό είναι λίγο περίεργο βέβαια γιατί εργάζεται κανείς σε μία γλώσσα με όλες τις αποχρώσεις, τις ρυθμίσεις, τις νομικές, τις ε, ρυθμίσεις, τις συντακτικές, τις επιπτώσεις τις κάθε λέξεις και ξαφνικά με τις μεταφράσεις χάνεις εντελώς τον έλεγχο βέβαια σε τόσες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά αυτή είναι και η ομορφιά, ο πλούτος της Ένωσης και θα πρέπει να ζήσουμε με αυτήν. Σχετικά τώρα με τη συγκεκριμένη έκθεση. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πιο απτές, αν θέλετε, τα πιο απτά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από αυτά είναι η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών στον χώρο Σέγγεν. και θα πρέπει το επίτευγμα αυτό να προσπαθήσουμε να το διατηρήσουμε. Θα πρέπει όμως να είμαστε και ειλικρινεί για το τι έχει συμβεί τους τελευταίους μήνες σχετικά με το δικαίωμα αυτό, το δικαίωμα να ταξιδεύει κανείς χωρίς να υφίσταται συνοριακούς ελέγχους εσωτερικού τύπου. Η αλήθεια είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια τα πράγματα πήγαν σχετικά καλά. Η επαναφορά ε, προσωρινών ελέγχων ε, έγινε δεκτή μόνο ε, κάποιες φορές, λίγες φορές, σε σχέση με πολύ μεγάλες απειλές οι οποίες είχαν εκφραστεί στα πλαίσια των εσωτερικών πολιτικών των κρατών μελών. Όμως, τους τελευταίους μήνες, τον τελευταίο χρόνο θα έλεγα, κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Κάποια πράγματα έχουν αλλάξει και ακριβώς αυτό μας οδήγησε στην συζήτηση εκ νέου της, ε, του δικαιώματος ελεύθερης διακίνησης. Όλοι θα ενθυμίστε ότι την προηγούμενη άνοιξη και στα πλαίσια της Αραβικής Άνοιξης ε, Ήρθαν πάρα πολλοί πρόσφυγες ε, στις ευρωπαϊκές ακτές και οι αντιδράσεις ορισμένων κρατών μελών ήταν στα όρια θα έλεγα της νομικής τάξης της σχετικής με τη Συμφωνία Σέγγεν. Η Ιταλία επέτρεψε σε αυτούς τους πρόσφυγες, ε, τους έδωσε τη δυνατότητα προσωρινά να παραμείνουν εκεί και να κυκλοφορήσουν. Ελεύθερα η Γαλλία όμως αποφάσισε μετά από αυτό να επαναφέρει τους συνοριακούς ελέγχους στα σύνορα με την Ιταλία. Σε εκείνη τη φάση ζήσαμε και μια μυστήρια πρωτοβουλία της ε, κυβέρνησης της Δανίας η οποία είπε ότι η επαναφορά των συνοριακών ελέγχων ήταν κάτι το οποίο χρειαζόταν η χώρα αυτή για να καταπολεμήσει το οργανωμένο έγκλημα. Μια αντίστοιχη περίεργη πρωτοβουλία πήραν οι Ολλανδικές αρχές με κάμερες οι οποίες τοποθετήθηκαν στα σύνορα και σε αυτή τη φάση η Επιτροπή έχει προχωρήσει στην ανάλυση του μέτρου. Και υπήρξαν και κάποιες άλλες πρωτοβουλίες που ακολούθησαν κάποια τραγικά γεγονότα όπως αυτά που συνέβησαν στην Νορβηγία. Η κυβέρνηση της Νορβηγίας σε εκείνη τη φάση αποφάσισε να επαναφέρει τους ε, συνοριακούς ελέγχους για λίγες ώρες ούτε καν μέρες. Πάντως, αυτά τα οποία συνέβησαν στα πλαίσια της ζώνης Σέγγεν, μας οδήγησαν στο να δούμε το θέμα αυτό με μεγαλύτερη προσοχή. Δεν ξέρω αν ενθυμίστε, πρέπει να ενθυμίστε. Είχαμε κάνει μία συζήτηση στην Ολομέλεια και μετά από τη συζήτηση αυτή είδαμε ότι δύο διαφορετικά θέματα τέθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ένα από το Συμβούλιο και το άλλο από το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρήσει με κάθε κόστος το κεκτημένο, το επίτευγμα το, στο οποίο έχουμε καταλήξει στον χώρο αυτό. Η Επιτροπή επανήλθε με μια συγκεκριμένη πρόταση σχετικά με την επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα κάτω από έκτακτες συνθήκες. Μια πρόταση η οποία ήταν πολύ ιδιαίτερα συμβατή θα έλεγα με αυτά τα οποία είχε ζητήσει το Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε την πρόταση που έκανε εκφράζοντας ξεκάθαρα τη βούλησή της να κρατήσει τη δυνατότητα λήψης απόφασης σχετικά με την επανεισαγωγή στα πλαίσια της επιτροπολογίας. Αυτή ήταν η νομική βάση. Η πρόταση αυτή αντιμετωπίστηκε με διαφορετικό τρόπο από τα διάφορα κράτη-μέλη από το Συμβούλιο και από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προσπαθούμε να είμαστε πραγματιστές, αποδεχόμεθα την πραγματικότητα δηλαδή και μπορεί εγώ προσωπικά να λέω ότι η πρόταση της Επιτροπής είναι πάρα πολύ καλή, και καινοτόμος, αλλά παρόλα αυτά αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα η πρόταση αυτή στο Συμβούλιο μέχρι τώρα. Λοιπόν, και εκφράστηκαν αρκετά επιχειρήματα από ορισμένα κράτη-μέλη. Με διαφορετικά επίπεδα αντίδρασης, αλλά πάντως υπήρξε διαφοροποίηση. Όταν κατέληξα λοιπόν στο φάκελο, Προσπάθησα να συνεισφέρω κι εγώ στα πλαίσια του κεκτημένου Σέγγεν, χωρίς φυσικά να το παίζω πόντιος πιλάτος και να λέω ότι όλοι έχουν δίκιο και όλοι θα προχωρήσουν με την άποψή τους. Επέμεινα ότι πρέπει να υπάρξει όμως μια κοινοτική διάσταση στην λήψη απόφασης για την επαναφορά ελέγχου. Χωρίς ίσως να προτείνω ακριβώς αυτό το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλαδή την επιτροπολογία. Γιατί όχι μόνο τα κράτη-μέλη εξέφρασαν την διαφορετική τους άποψη, αλλά και σε αυτήν εδώ την Επιτροπή όταν έγινε η πρώτη συζήτηση, πολλοί συνάδελφοι από πολλές πολιτικές ομάδες ξεκαθάρισαν ότι δεν θεωρούν η επιτροπολογία είναι ο σωστός τρόπος. Συνεπώς, αυτό το οποίο προτείνει σε αυτή τη φάση η έκθεση είναι το εξής. με έναν ιδιαίτερα συντονισμένο τρόπο όταν πρέπει να υπάρξει επαναφορά ελέγχου. Μέχρι τώρα προεβλέπεται ότι ένα κράτος μέλος όταν θεωρούσε ότι κάτι άλλαξε και επηρεάζει και απειλεί την εθνική του ασφάλεια ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόθεσή του να επαναφέρει τους συναδιακούς ελέγχους, ελέγχους, αλλά έχει πάντα τη δυνατότητα να λάβει την απόφαση. Η πρόταση που κάνω εγώ είναι να αλλάξει αυτή η κατάσταση κατά κάποιο τρόπο, λέγοντας ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα με πιο συντονισμένο τρόπο. Δηλαδή, όταν ένα κράτος μέλος, και αναφέρομαι σε προβλέψιμα συμβάντα βέβαια, όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι κάτι θα επηρεάσει την πολιτική του και την εθνική του ασφάλεια, μπορεί να ληφθεί απόφαση για επαναφορά ελέγχου σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με φυσικά την συνένεση της χώρας στην οποία, στις οποίες τα σύνορα θα επανέλθει ο έλεγχος. Τα κράτη-μέλη λοιπόν παραμένουν ουσιαστικά αυτά τα οποία λαμβάνουν τις αποφάσεις, αλλά όπως είπα, για να ληφθεί απόφαση θα πρέπει στο ίδιο τραπέζι να υπάρχει αντιπρόσωπος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της ομόρου χώρας. Στην περίπτωση μη προβλέψιμων συμβάντων, εκτάκτων καταστάσεων, η απόφαση φυσικά θα ληφθεί απόλυτα από τα κράτη-μέλη. Η διάρκεια του ελέγχου αυτού μπορεί να είναι κατά μέγιστον 10 ημέρες και μετά θα επαναληφθεί η διαδικασία αυτή την οποία είχα προβλέψει προηγουμένως τη παρουσία δηλαδή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της γειτονικής χώρας. Υπάρχει ένα θέμα, ένας τομέας και το βλέπει κανείς και σχετικά με την γλώσσα την οποία χρησιμοποιεί η έκθεση, η οποία δεν αναφέρεται μόνο στις δημόσιες πολιτικές και την απειλή στα θέματα ασφαλείας για μια χώρα, αλλά αναφέρεται επίσης σε έναν χώρο ο οποίος ε, χαρακτηρίζεται χώρος χωρίς εσωτερικά σύνορα και χωρίς συνοριακούς ελέγχους. Είναι αλήθεια ότι στην περιοχή Σέγγεν έχουμε μέλη τα οποία δεν είναι βέβαια μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πράγματα περιπλέκονται. Ταυτόχρονα είναι φυσιολογικό να πιστέψει κανείς ότι κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει μια χώρα ταυτόχρονα θα επηρεάσει το σύνολο της ζώνης Σέγγεν. Η μόνη κατάσταση στα πλαίσια της οποίας ε, ε, ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Επιτροπολογίας πράγματι θα είναι καθοριστικός είναι μια έκτακτη, πραγματικά έκτακτη κατάσταση, απρόβλεπτη, όπου υπάρχει σημαντική αδυναμία ελέγχου των εξωτερικών μας συνόρων. και αν ε, οι ανάγκες ε, δεν μπορούν να καλυφθούν με τον σωστό τρόπο, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποφασίσει την επανεισαγωγή των ελέγχων αλλά μόνο κάτω από πραγματικά έκτακτες συνθήκες όπου επιβεβαιούται μια έκτακτη ανάγκη αλλά υπάρχει αδυναμία κάλυψής της από τη χώρα μέλους. Λοιπόν, γιατί θέλουμε να αλλάξουμε τώρα την ισχύουσα κατάσταση. Κάποιοι πιστεύουν ότι τα πράγματα πήγαν καλά μέχρι τώρα. Γιατί θέλουμε να ανακατέψουμε τα χαρτιά και ίσως στο τέλος να καταστρέψουμε και κάτι το οποίο θεωρούμε ότι δουλεύει. Η απάντηση είναι ότι τους τελευταίους 12 μήνες κάποια πράγματα άλλαξαν. Όταν ένα κράτος μέλος λοιπόν φάνηκε ότι όταν ένας κράτος μέλος αποφασίζει να επανισάγει ε, τελωνιακούς ελέγχους, μεθοριακούς ελέγχους, δημιουργούνται ε, προβλήματα όταν η απόφαση λαμβάνεται μονομερός. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει θα έλεγα να ειδωθεί στα πλαίσια μιας τέτοιας κατάστασης σαν διαιτητής όταν υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σαν παράδειγμα. Εγώ συμφωνώ ότι εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι αυτή που θα αποφασίζει για την επαναφορά των ελέγχων. Τα κράτη-μέλη δεν θα θελήσουν να ενοχλήσουν το ένα το άλλο και γι' αυτό χρειαζόμαστε έναν αντικειμενικό διαιτητή θα έλεγα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένας τέτοιος δεν μπορεί παρά να είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να λάβει την κατάλληλη απόφαση. Τώρα, σχετικά με το ρόλο της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκφράσει επανειλημμένα την επιθυμία του να εμπλακεί ακόμα περισσότερο και να ενημερώνεται περισσότερο σε ό,τι έχει σχέση με τη ζώνη Σέγγεν για πολύ πρακτικούς λόγους το Κοινοβούλιο, ε, αυτή είναι η άποψή μου, δεν μπορεί να εμπλακεί στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων. Τα θέματα αυτά είναι θέματα τα οποία απαιτούν ένα κάποιο επίπεδο εμπειρογνωμοσύνης, όπως επίσης και μία κάποια ταχύτητα στον τρόπο λειτουργίας. Αυτό το οποίο προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι Τέσσερις εβδομάδες μετά από την ανέρεση των εσωτερικών ελέγχων το κράτος μέλος να έρχεται στο Κοινοβούλιο και να παρουσιάζει ε, μια αιτιολόγηση θα έλεγα και εξήγηση της επαναφοράς του ελέγχου. Και γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει η έκθεση να έρχεται σε αιτήσια βάση να συζητά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλες τις περιπτώσεις τις οποίες υπήρξε εισαγωγή ε, συνοριακών ελέγχων. Όπως επίσης και τις συνέπειες ε, της επανεισαγωγής αυτής και ταυτόχρονα και να υπάρξει και αξιολόγηση της ακρίβειας και της αναλογικότητας των μέτρων που λαμβάνονται. όλα με το θέλουν να παρεμποδίσουν. Εν ολίγης λοιπόν και θα σταματήσω για να ακούσω και τους συναδέλφους. και τα σχολιά τους. Αυτά είναι η λογική και τα επιχειρήματα που έχουν υπαγορεύσει την έκθεση αυτή. Περνάμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Νταπάκ, παρακαλώ. Εκ μέρους της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σε όλους. Θα αρχίσω επενθυμίζοντας την προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για το θέμα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να κρατήσει το πακέτο διαχείρισης Σέγγεν μαζί. Είναι εδώ και ο κύριος Κόλλιο. Και χαίρομαι που και η Προεδρία της Δανίας προσπαθεί να διασφαλίσει ότι η δουλειά που γίνεται όσον αφορά τον μηχανισμό αξιολόγησης ε, Σέγγεν και την τροποποίηση του κώδικα Σέγγεν είναι δύο πράγματα τα οποία τα βλέπει μαζί. Καλώς ορίζουμε λοιπόν την έκθεση της κυρίας Βέμπερ συμμερίστε τους στόχους της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι πρώτον να ενισχύσουμε τη διαχείριση του Σέγγεν με συντονισμένο πλαίσιο που να περιλαμβάνει εξαιρέσεις, κινδύνους, ειδικές περιπτώσεις. Δεύτερος στόχος είναι οι έκτακτες περιπτώσεις όπου πρέπει προσωρινά να επανισχύσουν οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα σε Πραγματικά όμως εξαιρετικές περιπτώσεις. Όπως σας είπα, μας ικανοποιεί πολύ το γεγονός ότι η έκθεση τονίζει ότι η μετανάσταση από μόνη της δεν πρέπει να θεωρείται ως απειλή στην ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πεπισμένη γι' αυτό και ξέρω ότι πολλοί το είπαν και στην προηγούμενη συνεδρία της Επιτροπής αυτής. Έρχομαι τώρα στις ειδικέ ε, περιπτώσεις, τις δύο ειδικέ περιπτώσεις που προβλέπονται ώστε εκτάκτος και προσωρινά να γίνεται επαναφορά των ελεγχών στα εσωτερικά σύνορα. Μερικές φορές βέβαια έχουμε πρόβλεπτες ε, ε, περιπτώσεις, συγκυρίες, όπως είναι αθλητικές ε, διοργανώσεις. Πρέπει όμως, όπως και μέχρι τώρα, να μπορεί το κράτος να αποφασίζει για ε, κατεξαίρεση επαναφορά των συνόρων για λόγους ασφάλειας. Το μηχανισμό αυτό βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτιμούσε να τον δίνει να ανατίθεται σε ένα ευρωπαϊκό κέντρο. Ε, ένα μηχανισμό κεντρικό που να αποφασίζει βάσει της επατροπολογίας. Παρ' όλα αυτά να γνωρίζουμε την ευαισθησία που έχει το κάθε κράτος μέλος όπως εκφράζει και η συγκίτρια. Γι' αυτό και μας ικανοποιεί ο τρόπος με τον οποίο λαμβάνει υπόψη στην ευαισθησία αυτή η συγκίτρια στην έκθεσή της και μιλάει για συντονισμένη προσέγγιση. Συνεπώς πρέπει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορούμε να ζυγίζουμε τα πράγματα και αναλογικά να λαμβάνονται οι αποφάσεις μόνο όταν αυτές είναι αναγκαίες, λαμβάνοντας υπόψη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Και όπως τονίζει η συγγήτρια, τα κράτη-μέλη ε, επηρεάζονται ε, άμεσα από τέτοιους ε, ελέγχους. Προτείνεται λοιπόν ισορροπία στην έκθεση και είναι κάτι που έχει συζητήσει και η ομάδα εργασίας στο Συμβούλιο υπό την Ιδανική Προεδρία. Όμω, και όπως είπα και τον προηγούμενο μήνα στη συνεδρίαση, πρέπει να εκφράσουμε ανησυχίε για την πρόταση που γίνεται στην έκθεση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να θετήσει κατευθυντήριε γραμμέ για την επαναφορά ε, των ε, ελέγχων για λόγους ασφάλειας. Αυτό αναφέρεται στην ε, τροπολογία 12 ως νομική υποχρέωση. Εμείς συμμεριζόμαστε την άποψη της εισηγήτριας για το ότι πρέπει να υπάρχει κάποια κατευθυντήρια γραμμή ώστε συνεκτικά να εφαρμόσετε το κεκτημένο Σέγγεν και αυτό το είπαμε και ήδη από το Σεπτέμβριο και ετοιμάζουμε κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι στα σύνορα αλλά και σχετικά με το θέμα των εγγράφων ε, των ταξιδιωτικών. Όμω, έχει αμφιβολίες για το κατά πόσο πρέπει να υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμέ για τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη-μέλη θα αξιολογούν ε, τις απειλέ στην ασφάλειά τους και τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στην ελεύθερη διακίνηση. Τέτοιε αξιολογήσεις πρέπει να γίνονται κατά περίπτωση, ε, συχνά βάσει πληροφοριών ιδιαίτερα ευαίσθητων, μυστικών πληροφοριών πολλές φορές. Πρέπει να Είμαστε αποτελεσματικοί και ξέρω ότι δεν θα συμφωνήσω το κρατημέλη με κάτι τέτοιο. Πάντως, η ύπαρξη μιας τέτοιας απειλής, βάση δηλαδή εθνικής πολιτικής ή ασφάλειας, δεν είναι κάτι που αρκεί για να επανέλθουν οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα. Γι' αυτό και υπάρχει το νέο άρθρο 23α που προτείνουμε δηλαδή, που ζητάει μια επιπλέον δοκιμή να γίνεται για να δούμε κατά πόσο τηρείται η αναλογικότητα ή όχι. Υπάρχουν κάποιες έκτακτες περιπτώσεις όπου η επανεισαγωγή των ε, ε, ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα μπορεί να επιβάλλεται εφόσον υπάρχουν ελλείψεις για παράδειγμα. Πάντως, χαιρόμαστε που αναφέρεται η ανάγκη για μηχανισμούς στο νέο άρθρο 26 που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε έκτακτες συνθήκες και ως ίστατη λύση να μπορεί να είναι η επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Πιο πολύ πρέπει να δούμε ε, πόσο τηρούνται οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως αναγνωρίζουμε ότι μια τέτοια απόφαση επαναφοράς πρέπει να λαμβάνεται συντονισμένα κατά προτίμηση μέσω της επιτροπολογίας. Τέλος, επιτρέψτε μου να σας πω κάτι και για την πρόταση που γίνεται στην έκθεση για την αναφορά. Η Επιτροπή συμμερίζεται την άποψη ότι πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και λογοδοσία όσον αφορά την διαχείριση του χώρου Σέγγεν και ότι κάτι τέτοιο βελτιώνεται μέσω ενισχυμένου διαλόγου ανάμεσα στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο βάσει ειδικών αναφορών που θα γίνονται από τα κράτη-μέλη αλλά και τακτικών αναφορών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως γνωρίζετε, στην ανακοίνωσή μας το Σεπτέμβριο που μας πέρασε αναφέρουμε ετήσια εκθέση, μάλλον δύο φορές το χρόνο όσον αφορά τη λειτουργία του Σέγγεν και η πρώτη τέτοια έκθεση θα γίνει στα τέλη του Μαΐου φέτος. Σίγουρα θα είναι εφικτό μία φορά το χρόνο, κάθε δεύτερη αναφορά που κάνουμε, να έχουμε και μία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία να λαμβάνει υπόψη την ε, εμπειρία που έχουμε όσον αφορά τις ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα κάθε φορά που έχουν ε, αυτά επανέλθει κατά την ε, τελευταία χρονιά. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το σύστημα διαχείρισης Σέγγεν σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό. Ευχαριστώ. Η Προεδρία τώρα, λέει ο Πρόεδρος, <clears throat> θέλει να πει κάτι, μήπως ε, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Η Προεδρία θέλει να ευχαριστήσει την κυρία Βέμπερ για την, ε, το σχέδιο έκθεσής της που μας προτείνει. Πιστεύουμε ότι το σχέδιο έκθεσης όντως αποτελεί μια πολύ καλή βάση για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις. Θέλουμε επίσης να ενημερώσουμε τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ ότι με την πρόταση αυτή και με την έκθεση για το μηχανισμό ΣΕΒΑΛ ε, είναι αντικείμενο εργασίας στην ομάδα εργασίας μας και συνεχίζει η δουλειά δηλαδή πάνω σε αυτά τα δύο θέματα. Θα υπάρξουν και διαπραγματεύσει βέβαια με το Κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Είναι αναγκαίο να λάβουμε υπόψη μας ότι θέματα τα οποία έχουν με την δημόσια τάξη και την εσωτερική ασφάλεια και ιδιαίτερα με τους ελέγχους στα σύνορα είναι θεμελιώδη. Τα κράτη-μέλη, όπως υπογραμμίζει το Συμβούλιο, ε, πιστεύουν ότι η ασφάλεια των ατόμων, μάλλον ότι η ελεύθερη διακίνηση των ατόμων είναι ένα μεγάλο επίτευγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Σέγγεν και γι' αυτό το σύστημα αυτό πρέπει να παραμείνει. Τέλος, Θέλουμε για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια και να ευχαριστήσουμε και όλα τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για την καλή συνεργασία που είχαμε μαζί τους. Προσδοκούμε σε έναν επικοδομητικό διάλογο στο μέλλον. Ευχαριστώ. Οι σκιώδεις μας τώρα. Με τον κύριο Κόγιο πρώτο. Θέλετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ξεκινώντας θα ήθελα να ευχαριστώ τη Ρενάτα Βέμπερ για την έκθεση. Και να επισημάνω σε όλους του συναδέλφου ότι είναι ξεκάθαρο πω η Ρενάτε προσπάθησε, να, προσπάθησε πολύ να εξασφαλίσει ε, συνετική συμβιβαστική θέση ως προς προτάσεις του Συμβουλίου. Χαίρομαι γιατί βλέπω ότι έχουμε τις ίδιες κοινέ γραμμές, τις ίδιες κοινέ κόκκινες γραμμές που πρέπει να προσδορίζουν τις θέσεις του Κοινοβουλίου και τη διακυβέρνηση Σέγγεν. Πρώτο σημείο. Η Ρενάτα ξεκάθαρα υποστηρίζει την ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέος μηχανισμός Σέγγεν, ο οποίος θα εξασφαλίζει την σαφή και συνεπή εφαρμογή του κεκτημένου και Σέγγεν. Δηλαδή, η τελωνιακή ή η συνοριακή έλεγχη θα πρέπει να αποτελέσουν μια εξέλιξη, μια συνέπεια της εξέλιξης του Σέγγεν και όχι νέα προσχήματα για επαναφορά των ελέγχων στην Ευρώπη. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο να ενισχυθεί η ασφάλεια, αλλά και να ενισχυθεί η ελεύθερη διακίνηση των πολιτών, να ενισχυθούν τα δικαιώματα των πολιτών και να παρακολουθείται με πολύ μεγάλη προσοχή οδήποτε απόπειρα για επαναφορά ελέγχου στα ιστορικά σύνορα, έστω και νομίμων, με το πρόσημα τη νομιμότητα. κάποιε προσπάθειε πρόσφατε των ε, κρατών μελών, ορισμένων κρατών μελών, εξηγούν γιατί πρέπει να το πράξουμε αυτό. Πρέπει να καθισχάσουμε του πολίτε μα ότι νέα μέτρα λαμβάνονται προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα όπως αυτά που έχουν να κάνουν με την, όπως αυτά που οδηγούν σε παραβίαση κυριότητας και περιορισμό των, δικαιωμάτων στον χώρο Σέγγεν. Τέλος. Είναι πολύ σαφές ότι Ρενάτε ξεκάθαρα υπογραμμίζει τη σημασία των μεταναστευτικών ροών, οι οποίες αυτές καθεαυτές δεν μπορούν να θεωρηθούν ως απειλή και απευθείας λόγος εισαγωγής ε, συνοριακών ελέγχων. Εφόσον τηρηθούν αυτές οι κόκκινες γραμμές, πιστεύω θα μπορέσουμε να βρούμε μια καλή λύση. Υπάρχουν κάποιοι, κάποια περιθώρια βελτίωσης φαντάζομαι και διαβεβαίνω τη Ρενάτε ότι θα καταθέσουμε τις τροπολογίες μας στη Ρενάτε όταν έχουμε τη δυνατότητα, το χειρότερο δυνατό. Ευχαριστώ πολύ και εσείς, κύριε Ένσου, που ήσασταν επίσης σκιώδης. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εδώ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όλες σχεδόν οι πολιτικές ομάδες έχουν την ίδια άποψη για το θέμα αυτό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σε μια δύσκολη στιγμή, όπως τώρα, καθώς το Συμβούλιο ε, αρνείται να διαπραγματευτεί την πρόταση αυτή από την Επιτροπή, βρισκόμαστε λοιπόν σε μια δύσκολη κατάσταση, δεδομένου ότι τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο, που είναι εκείνα τα οποία είχαν ζητήσει έναν τέτοιο μηχανισμό, τώρα θεωρούν ότι δεν τα εκφράζει πλέον, ότι δεν έχουν σχέση με την υπόθεση αυτή. Και έτσι, όπως είπε και ο Σάνφο νωρίτερα, πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποιε προτεραιότητες. Καταρχάς, οι προτεραιότητες. Στο Συμβούλιο. Περιμένω από την Προεδρία της Δανίας να συμβάλλει στην ε, βελτίωση της τάσης του Συμβουλίου, ώστε να ξεβρεθεί μια επικοδομητική λύση. Δεύτερον, δεν πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ανησυχήσει από την άρνηση του Συμβουλίου και όπως είπαν και οι συνάδελφοι μπορούμε να προσδιορίσουμε ήδη μια προκαταρκτική απόφαση για ένα μηχανισμό διαφύλαξης, ένα συντηρητικό μηχανισμό, ο οποίος ε, θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρώτο μήνυμα προς τα κρατη Και πάντως πρέπει να έχουμε σε σημείο κίνησης ότι η ελευθερία της διακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών είναι δεδομένη και ότι οι έλεγχοι στα σύνορα, στα ιστορικά σύνορα μπορούν να επανέρχονται μόνο σε άκρος εξαιρετικές περιπτώσεις. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι τώρα, οι μεταναστευτικές ροές δεν πρέπει να αποτελούν απειλή για τη δημόσια ασφάλεια. Οι πάντε συμφωνούν για το γεγονός, το γεγονός αυτό. Και είπαμε ότι ο μηχανισμός ε, θα πρέπει να είναι κοινοτικό μηχανισμός και όχι μηχανισμός ο οποίος θα εξαρτάται από το κάθε κράτος μέλος. Από την άλλη μπορούμε να διαπραγματευτούμε συγκεκριμένες πτυχές της υπόθεσης, καθώς το Συμβούλιο λοιπόν αντιτάσσεται στην πρόταση αυτή της Επιτροπής. Δεν ξέρω αν η επιτροπολογία μπορεί να αποτελέσει την καλύτερη λύση. Νομίζω ότι θα πρέπει πάνω απ' όλα να ξεβρεθεί μια πιο διαφανή λύση που θα επιτρέψει εμά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με το Συμβούλιο και την Επιτροπή, να ε, λάβουμε αποφάσει σημαντικέ πάντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εν τέλει, μεγάλη σημασία και θεμελιώδη έχει το εξή ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται για κάθε απόφαση που λαμβάνεται σε σχέση με, την, τον χώρο Σέγγεν. Είναι πολύ σημαντικό για τον Ευρωπαίο πολίτη να να έχει την να εκπροσωπείται στις ε, διαδικασίες αυτές και ελπίζω ότι η κυρία Βέμπερ θα δέχεται τις προτάσεις αυτές ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις... Ελπίζω το Συμβούλιο θα δέχεται τις προτάσεις κυρία Σέγγεν ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την έγκριση του πακέτου αυτού. Είναι σαφές ότι ο μηχανισμός αξιολόγησης για το χώρο Σέγγεν έχει επίσης μεγάλη σημασία. για την τηρήση του στόχου διακυβέρνησης το χώρο Σέγγεν. Ευχαριστώ την κυρία Σέγγεν, την κυρία Βέμπερ. Και πάνω απ' όλα, πάνω για τις εξαιρετικές της ικανότητες, τις διαπραγματευτικές, για τη βούλησή της να ε, απεμπλέξει την διαδικασία λήψη αποφάσης στην υπόθεση αυτή από, τις, τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τανακή Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να εκφράσω την ελπίδα πως οι διαπραγματεύσεις αυτές στο Συμβούλιο θα οδηγήσουν σε μια σωστή λύση. Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση. Έχουν εκφραστεί τα επιχειρήματα από τους συναδέλφους. Δεν θα τα επαναλάβω. Πλην όμως, για την κυρία Βέμπερ, τι θέλω να πω. ότι ναι, έχετε πολλή δουλειά μπροστά σας ακόμη για τις διαπραγματεύσει. Η θέση μας πάντως στις διαπραγματεύσει αυτές θα μπορούσε πιστεύουμε να είναι πολύ πιο σκληρή, να ακολουθήσουμε πιο σκληρή γραμμή. πιστεύουμε ότι η πρόταση για την επανεισαγωγή μέτρων ε, των 10 ωρών που αναφέρεται σε εξαιρετικέ περιπτώσεις είναι υπερβολικά ε, μεγάλη περίοδος και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μία παράταση που φτάνει μέχρι τους δύο μήνες. Δεν ξέρω με καταλαβαίνεις Ρενάτη έτσι όπως μιλάω ή αν καταλαβαίνεις εσύ το, τις θέσεις του Συμβουλίου καλύτερα. Πάντως η ομάδα μας θεωρεί ότι οι χρονικές περίοδοι που προτείνονται είναι μεγάλες και θα έπρεπε να συντομεύσουν πέντε μέρες ίσως για την εισαγωγή. Επίσης, με ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι η συγγήτρια πιστεύει ότι οι μεταναστευτικές ροές δεν μπορούν αυτές αυτές να θεωρηθούν ως κίνδυνος για την εσωτερική ασφάλεια Και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί ένα συγκεκριμένο ορισμό του τι συνιστά δημόσια ασφάλεια ή απειλή για τη δημόσια ασφάλεια και την εσωτερική τάξη με πολύ αυστηρή διατύπωση. Συμφωνούν οι συνάδελφοι, συμφωνεί η συγγήτρια, όπως και εμείς, ότι ο ορισμό αυτός δεν μπορεί να περιλαμβάνει αναφορά σε μεταναστευτικές ροέ χωρί περαιτέρω διευκρίνηση. Επίσης πιστεύουμε ότι προβλήματα σχετικά με εσωτερικές διαδικασίες δεν μπορούν να αποτελέσουν λόγω επανεισαγωγής ελέγχων στα ιστορικά σύνορα. Αυτή είναι η θέση μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι δύσκολες πραγματεύσεις, όπως ακούστηκε Ελπίζουμε ωστόσο ότι η Προεδρία της Δανίας, όπως άλλωστε μας είπε, θα κάνει ό,τι μπορεί για να καταλήξουμε σε μια καλή συμβαστική λύση. Σας ευχαριστώ. Κυρία Μάκιντσάια. Ευχαριστώ. Εν γέννη, η ομάδα μας τίνει να δείχνει κατανόηση στις ανησυχίες των κρατών μελών και θεωρούμε ότι έχουν εύλογες ανησυχίες και σωστά ζητούν κάποιες ασφαλιστικές επιπτώσεις προς την ε, εσωτερική ασφάλεια. Βέβαια, εν γέννη επίσης έχουμε, τρέφουμε ιδιαίτερη εκτίμηση για τη δουλειά και τις προσπάθειες της κυρίας Βέμπερ στην υπόθεση αυτή. Πιστεύω ότι θα μπορέσει να φέρει την έκθεση σε ένα καλό σημείο. Έχω μια ερώτηση. Καθώς βρίσκομαι σε πλεονεκτικότερη θέση, μια και τα αγγλικά είναι μετρική μου γλώσσα και ξέρω ότι δεν έχει μεταφραστεί στις λοιπές η έκθεση αυτή. Σημειώνω πάντως ότι η πρόταση της Επιτροπής, στις προτάσεις της Επιτροπής, χρησιμοποιείται η έννοια Common Union Response, κοινή ενωσιακή ανταποκρίση. Ενώ σε άλλα σημεία αναφέρεται μόνο η έννοια Common Response. Ποια είναι η διαφορά και η κυρία Βέμπερ πώς την αξιολογεί. Ε, για δε την Προεδρία και έχοντας υπόψη τις αντιδράσεις των κρατών μελών, τις τοποθετήσεις τους. Σας ερωτώ λοιπόν εσείς πώς κρίνετε τις πιθανότητες να εγκριθεί τελικά το θέμα αυτό, να καταλήξουμε σε συμφωνία δηλαδή. Κυρία Ernst, ο Σκιώδης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστώ την εισηγήτρια, την κυρία Βέμπερ. Ξέρουμε, έχει πολύ καυτά κάρβουνα να βγάλει από τη φωτιά. Και πάνω απ' όλα έχει να κάνει με ένα πλαίσιο πολύ αυστηρών προδιαγραφών θα πρέπει να εισαχθούν εάν πρόκειται να περιστέλλεται η ελεύθερη διακίνηση ή να επανισάγονται έλεγχοι στα σύνορα. Όλα αυτά τα λέω διότι δεν πιστεύουμε ως ομάδα απολύτως ότι χρειάζεται ένας τελείως νέος μηχανισμός και ως εκ τις προσπάθειές μας θα τις κατευθύνουμε περισσότερο προς την ενίσχυση προς την ε, προσπάθεια καλύτερα να αποφευκθεί όσο το δυνατόν, να περιορίζεται δηλαδή και να είναι όσο το δυνατόν πιο αυστηρή η όρη για την υπανεισαγωγή αυτών των ελέγχων στα σύνορα. Πιστεύω ότι κύριε, με την κυρία Βέμπερ θα έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Ε, δεύτερο σημείο, πιστεύουμε ακράτατα στην κοινοτική μέθοδο, ειδικά όταν πρόκειται για, με, για αποφάσεις που έχουν να κάνουν με την επανεσταγωγή των ελέγχων στα ιστορικά σύνορα Φερρυπίν. Και για να έχουμε και ασφάλεια βεβαίως ε, δικαίου αλλά και διαφύλαξη της ελεύθερης διακίνησης των πολιτών πρέπει η κοινοτική μέθοδος να είναι εκείνη η οποία θα καθορίσει ή μη τι άλλο θα έχει το καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση αυτή. Από την άλλη, κάποιες ε, ανησυχίες εκφράζοντας προς το κατά πόσον ε, μπορεί για τα κράτη-μέλη να αφαιθούν ανοιχτά παραθυράκια στο νομοθέτημα, τα οποία θα τους επέτρεπαν να ε, καταστρατηγούν τις ε, αυστηρές διατάξεις. Θα πρέπει να τα κοιτάξουμε αυτά με πολύ μεγάλη προσοχή. Και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι εξάπαντος πρέπει να παραμείνει η ο αποκλεισμό της μετανάστευσης ως αυτής καθεαυτής ως κριτηρίου απειλής της δημόσιας ε, ασφάλειας, της ιστορικής ασφάλειας. Αυτό οπωσδήποτε πρέπει να παραμείνει όπως έχει. Δεν μπορεί να εισαχθεί δηλαδή και κυρίως ανεφετέρου ε, ως κριτήριο απειλής η μετανάστευση, μεταναστευτικές ροές. Θα θέλαμε πολύ πολύ σαφείς κανόνες δηλαδή, οι οποίοι με πολύ αυστηρούς όρους θα ε, επιτρέπουν πότε μπορεί να επανέλθει ο έλεγχος στα ιστορικά σύνορα με συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για τις 10 ημέρες η κυρία συνάδελφος από τους Πρασίνους είπε επίση ότι παρά είναι χαλαρό το χρονικό αυτό διάστημα, χρειάζεται πιο αυστηρή διάταξη, ίσως τρεις ημέρες ακόμη αντί για 10. Και πριν τελειώσω θα ήθελα να αναφερθώ στους ποσοτικούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα. Είναι κάτι το οποίο συζητούμε τακτικά. Τι σημαίνουν ποσοτικοί έλεγχοι, τι στόχο έχουν, τι σημαίνει ποσοτικός έλεγχος. Θέλουμε να το έχουμε λοιπόν απόλυτα ξεκάθαρο ώστε να μην υπονοείται μέσω των ποσοτικών ελέγχων για άλλη μια φορά ότι βάλουμε κατά τον μεταναστευτικών ροών. Προσπαθούμε να ε, αντιμετωπίσουμε με τον τρόπο αυτό τις μεταναστευτικές ροέ. Εν γέννη, λοιπόν, θα θέλω να πω ότι η έκθεση μα έχει κάνει καλή εντύπωση, αλλά βέβαια δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική και έτσι θα πρέπει να καταθέσουμε πλευρά τη ομάδα μα τροπολογίε. Ευχαριστώ. Δία Δεμήρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω διάφορα σχόλια σε σχέση με την έκθεση αυτή. Το πρώτο που θέλω να πω είναι τι είναι κοινό. Η δυνατότητα εργασίας και σίγουρα η Ρενάτε Βέμπερ είναι πολύ καλά εξοπλισμένη για να ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Ποιες είναι οι παρατηρήσεις μου τώρα. Πράγματι, θέλουμε να διαφυλάξουμε την ελεύθερη κυκλοφορία. Εφόσον κυκλοφορούν ελεύθερα τα κεφάλαια, οι υπηρεσίες, οι... τα εμπορεύματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε την ελεύθερη κυκλοφορία και των ατόμων. Δεύτερον, εφόσον όλα έχουν ρυθμιστεί και προβλεφθεί για αλλαγέ. Τι θέλουμε να αλλάξουμε, τι θέλουμε να ρυθμίσουμε, επειδή κάποιες χώρες πέρασαν αυτό που ονομάζουμε κόκκινες γραμμές. Όμως κάθε φορά που οι χώρες αυτές, που ξέρουμε πολύ καλά ποιες είναι, Κάθε φορά λοιπόν που περνάνε τις κόκκινες γραμμές υπάρχει μια αντίδραση ισχυρή. Και εμείς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης αντιδράσαμε. Όμως, όταν η κατάσταση είναι απρόβλεπτη, μάλλον όταν δεν είναι απρόβλεπτη, αλλά είναι μια αντίδραση απόλυτα δικαιολογημένη, τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και γενικά η Ευρωπαϊκή Κοινωνία δεν ε, αντιδράει. Και σε τι αναφέρομαι, θα σας πω αμέσω. 11η Μαρτίου, η επίθεση δηλαδή στις ε, 11η Μαρτίου στην Ισπανία ή και εκείνη που είχαμε πιο πρόσφατα στην Νορβηγία, όπου για ένα μικρό χρονικό διάστημα ε, επανέρχονται οι έλεγχοι στα σύνορα, τότε δεν αντέδρασε κανείς. Και γιατί, γιατί ήταν απόλυτα δικαιολογημένο. Όταν υπάρχει λοιπόν αιτιολόγηση, εντάξει, δεν είναι όμως αιτιολογημένο να ε, αναφέρει κανείς τους ελέγχους στα σύνορα επειδή υπάρχει μια μετανάστευση. Έχουμε πολλά παραδείγματα. Έχουμε η χώρα μου για παράδειγμα το 2006 από τον Ατλαντικό είχε τεράστια πίεση από τις μεταναστευτικές ροές. Δεν επανέφερε όμως τους ελέγχους στα σύνορα. Αυτό λοιπόν πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, η έκθεση αυτή δεν είναι αναγκαία, γιατί τι προσπαθεί να κάνει, να ρυθμίσει κάτι που είναι ήδη ρυθμισμένο. Το θέμα είναι τι κάνουμε όταν κάποιες χώρες δεν τηρούν τα όσα έχουν ήδη ρυθμιστεί και αποφασιστεί. Αυτό θα έπρεπε να είναι η ουσία της έκθεσης. Πάντως, με ή χωρίς ρύθμιση, νέα, οι χώρες που παραβιάζουν τις αρχές μας συνεχίζουν να το κάνουν. Διότι δεν προβλέπεται ε, κάτι στο κεκτημένο Σέγγεν για τις έκτακτες περιπτώσεις τι είναι το προβλεπόμενο, ας πούμε, μια αθλητική διοργάνωση. Αυτό μπορεί κανείς να ρυθμιστεί. Μπορεί να ενημερωθεί το Συμβούλιο, η Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, οι χώρες μέλη. Αλλά όταν έχουμε κάτι το απρόβλεπτο και κάποιος αντιδρά ε, αμέσως, αυτό πρέπει να συμβαίνει μόνο από μονομερός από τη χώρα μέλος η οποία εμπλέκεται για να μπορεί αποτελεσματικά να προχωρήσει σε έρευνες και σε δίωξη ενδεχομένω, σε περίπτωση απρόβλεπτου γεγονός, έτσι, γεγονότος, έτσι. Και μετά, βέβαια, να ενημερώνει και το Συμβούλιο και την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο. Αυτή είναι η άποψή μου, Πρόεδρε. Όταν έχω την μετάφραση της έκθεσης αυτή στην γλώσσα μου θα επανέλθω. Πάντως υπενθυμίζω ότι είχε πει το Κοινοβούλιο. Είπε το Κοινοβούλιο ότι εφόσον αυτό το θέμα έχει ρυθμιστεί, γιατί πρέπει να επανέλθουμε και να το ρυθμίσουμε και πάλι. Δεν θέλουμε ένα νέο και εκτιμένο, θέλουμε να τηρείται το ήδη υπάρχον και ισχύον. Ευχαριστώ κύριε Ρωμέρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτή τη φορά θα συμφωνήσω απόλυτα με τόσα μόλις είπε ο κύριος Δεμέρα. Και δεν ξέρω γιατί. Γιατί είμαστε και οι δύο Ισπανοί, Γιατί είδαμε και οι δύο τις μαζικές μεταναστευτικέ ροές που φτάσανε στη χώρα μας. Που δεν αναγκάσαμε ποτέ καμιά άλλη χώρα να περάσει ελέγχου για να μπει στη χώρα μας. Είναι γι' αυτό ή είναι γιατί είμαστε ρεαλιστέ σε αυτό το θέμα. Πάση περιπτώσει έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα πάνω στο οποίο όλοι συμφωνούν ότι ο στόχος, το αντικείμενο δεν μπορεί να είναι μεταναστευτικές ροές. Και όλοι γνωρίζουμε ότι ο κανονισμό αυτός είναι μια αντίδραση στο φαινόμενο της Λαμπεντούσα. Η Επίτροπος Μάλστρομ μας το παρουσιάζει σαν απάντηση ε, στην Λαμπεντούσα, δηλαδή μεταναστευτικές ροές. Μα στην ουσία έχουμε να κάνουμε εδώ με μια πρόταση που κατά τη γνώμη μας δεν θα έπρεπε να είναι απάντηση στις μεταναστευτικές ροές ε, που έφτασαν στη Λαμπεντούσα. Αλλά αν δεν είναι γι' αυτό, τότε γιατί, σε τι απαντάει. Δεν αιτιολογείται, δεν δικαιολογείται. Ακόμα και στην αιτιολογική σκέψη που αναφέρονται ε, το Σέγγεν, πώς δημιουργήθηκε, τι διαφορές υπάρχουν. Υπάρχει οδηγία του 2001 που μπορεί να πρέπει να αλλάξει, μπορεί ίσως αυτό να είναι απάντηση για τις περιπτώσεις που εξετάζουμε. Αλλά δεν πρόκειται εδώ για μια απάντηση στις μεταναστευτικές ροές. Γιατί δεν προτείνεται καν τροποποίηση της οδηγίας αυτής. Αυτό που έχει γίνει είναι ότι, όπω πολύ σωστά είπε ο κύριο δύο χώρε μέλη δεν τήρησαν τη συνθήκη. Δεν τήρησαν τις οδηγίες. Και η επίτροπο Μάλστρομ, ή τέλο πάντων Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αντί να επιστήσει την προσοχή μας σε αυτές τις χώρες και να πει σε αυτές τις χώρες παραβιάζετε την νομοθεσία, ενώ πρέπει να την τηρείτε, ήρθαν και μας έφεραν αυτόν τον κανονισμό. Ειλικρινά πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε και εμείς σοβαροί. Γιατί αν δουλέψουμε για να αντιμετωπίσουμε τις μεταναστευτικές ροές στη Λαμπεντούσα, ε, ας το κάνουμε, αλλά τότε να τροποποιήσουμε την οδηγία του 2001 ή ακόμα και στην έκθεση Παπα-Νικολάου. Γιατί όταν υπάρχει μια μεταρρύθμιση του Σέγγεν μπορεί να προβλέψουμε έκτακτες περιπτώσεις. Μπορεί να είναι στη γραμμή της τροπολογίας της κυρίας Μακοβέη με την οποία δεν συμφωνώ βέβαια, γιατί συνδέονται τα θέματα βλέπετε. Η ουσία είναι τι αποτελεί απειλή για την εσωτερική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη. Διότι ένα αθλητικό γεγονός αποτελεί απειλή για τη δημόσια τάξη και την ε, ασφάλεια, όπως πολύ σωστά λέει ο κύριος Δεμέρμα, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, γιατί δεν είναι όλες οι αθλητικές ε, διοργανώσεις απειλή. Πώς μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό, πώς μπορούμε να το ξέρουμε. Το θέμα της Νορβηγίας που επανέρχεται είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πραγματικά η Νορβηγία είναι μια απειλή. Δηλαδή η τρομοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί απειλή. Αλλά τότε δεν βοηθάει σε τίποτα όταν λέει ότι από πριν θα πρέπει να ενημερωθούν κτλ. Δεν έχει κανένα νόημα. Λέει 30 μέρες. Γιατί 30 μέρες και γιατί όχι 45 και γιατί όχι 60 αν η κατάσταση είναι έκτακτη, είναι έκτακτη. Ο κανονισμός αυτός δεν βοηθάει σε τίποτα σε περίπτωση τέτοιων έκτακτων περιστάσεων. Γι' αυτό και αυτά τα είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάποια στιγμή. Δεν μας βοηθάει σε τίποτα, δεν μας ε, ε, βοηθάει καθόλου σε έκτακτες περιπτώσεις ο κανονισμός αυτός. Και θέλω να πω στην κυρία Βέμπερη, η οποία έχει κάνει βέβαια τεράστια προσπάθεια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι είναι θεματοφύλακας των συνθηκών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν δεν μπορεί να δώσει κατευθυντήριες γραμμές, γιατί οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής είναι οδηγίε, οδηγίες. Τις οδηγίες πρέπει να τηρούμε, τη συνθήκη. Και έχει δίκιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία θα φτιάξει ένα πλαίσιο εκτός των οδηγιών της. Πράγματι λοιπόν πρέπει να προσπαθούμε να βρούμε μια απάντηση στο πρόβλημα της Λαμπαντούσα, αλλά δεν είναι ο κανονισμός αυτός όπως πολύ σωστά λέει και ο κύριο Κοέγιο, εντάξει, να αξιολογήσουμε, αλλά είναι το Σέγγεν που είναι η απάντηση έτσι καλλιώς ε, στα θέματα που συζητάμε. Πρέπει να ενισχύσουμε το σύστημα σύλλου, πρέπει να ενισχύσουμε του συνοροφύλακε. ό,τι πρέπει να ενισχύσουμε, να το ενισχύσουμε και ακόμα περισσότερο όταν υπάρχει έκτακτη ε, κατάσταση. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι επειδή θα υπάρξει κάποιο αθλητικό γεγονός, μια αθλητική διοργάνωση, εμείς θα φτιάξουμε αυτόν τον κανονισμό, μήπως και. Μα δεν είναι γι' αυτό. Εγώ λοιπόν συμφωνώ Δεν ξέρω το Συμβούλιο γιατί το κάνει αυτό, αλλά μπορώ να υποθέσω ότι είναι για να προστατευτούν οι χώρες οι οποίες δεν τήρησαν τις συνθήκες, τις οδηγίες που προβλέπονται για αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά δεν μπορεί εμείς να φτιάξουμε έναν κανονισμό για τον κύριο Σαρκοζή, για παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν. Εμείς είμαστε ένα σοβαρό κοινοβούλιο. Νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε τι θα κάνουμε και με όλη την καλή θέληση που έχει η κυρία Βέβερ, ειλικρινά, αυτό που κάνουμε τώρα δεν έχει καμιά σχέση με την ενίσχυση της διαχείρισης του Σέγγεν. Ο κανονισμός αυτός θα είναι στην πράξη άχρηστος. Μου δίνει την εντύπωση ότι χάνουμε το χρόνο μας με τον κανονισμό αυτό, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντέδρασε τότε που έπρεπε να αντιδράσει με τον τρόπο που έπρεπε να αντιδράσει. Ευχαριστούμε. Ε, <clears throat> κυρία Ματιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, μετά από αυτά τα οποία άκουσα δεν έχω πολλά να πω. Εγώ έχω ήδη συγχαρεί την κυρία Βέμπερ για την προσπάθεια που έκανε και για τη συμβιβαστική λύση στην οποία κατέληξε, γιατί το θέμα είναι πράγματι περίπλοκο. Αλλά θα συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες. Αν δει κανεί τι έχει γίνει από το 2006, κοινοποιήθηκαν 27 μόνο αποφάσεις επανεισαγωγής προσωρινών ελέγχων για σωστούς λόγους η Πορτογαλία σαν παράδειγμα για τη συνάντηση κορυφής του ΝΑΤΟ, για το φόρουμ το οικονομικό το παγκόσμιο στη Βιέννη, για την Ορβηγία για το λυπηρό γεγονός που γνωρίζουμε. Δεν θα σας αναφέρω όλες τις λεπτομέρειες. Και η Γαλλία, στην οποία αναφερθήκαμε ήδη σήμερα, την προηγούμενη άνοιξη, ε, για τη λεγόμενη Αραβική Άνοιξη. Δεν θα επαναλάβω λοιπόν αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, μίλησαν πάρα πολύ σωστά. Αλλά αν ήθελα να υπογραμμίσω ακόμα περισσότερο την κατάσταση θα έλεγα ότι αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε καταδικάσει και την Ιταλία για όλες αυτές τις άδειε αμφιβόλου χρησιμότητας τις οποίες είχε διανύμει στους ξένους και επίσης είχε καταδικάσει και τη Γαλλία για την επαναφορά αυτή τη μονομερή των ελέγχων τότε δεν ε, θα χρειαζόταν να γίνει όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται σήμερα και από την κυρία Βέμπερ. Εν πάση περιπτώσει η πρόταση που έχουμε εδώ μπροστά μας σήμερα δεν βοηθάει σε τίποτα την κατάσταση και νομίζω ότι μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση, δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Πίρκερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι υπάρχει ουσιαστικά ομοφωνία γύρω από την αξιολόγηση του μηχανισμού Σέγγεν. Νομίζω ότι όλοι βλέπουμε θετικά τη ζώνη Σέγγεν. Νομίζω ότι η ζώνη Σέγγεν είναι ε, υπόδειγμα αποτελεσματικότητας και σωστής πειθαρχίας και καλώς εννοούμενης πειθαρχίας. Επίσης όλοι θα συμφωνήσουμε ότι μόνο στην περίπτωση κατά την οποία απειλείται η ασφάλεια μιας χώρας τότε θα πρέπει να έχει το δικαίωμα μονομερούς επαναφοράς εσωτερικών ελέγχων. Συνεπώς όταν διαπιστούνται μια τέτοια απειλή είναι φυσιολογικό μια χώρα να ζητήσει την επαναφορά των εσωτερικών ελέγχων για μια συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Συγγνώμη για το τηλέφωνο μου που χτύπησε δίπλα από το μικρόφωνο. Λοιπόν βλέπουμε λόγω κάποιων πρόσφατων συμβάντων ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν πάντα όπως εμείς τα θέλαμε να πηγαίνουν. Δεν ζούμε σε ένα ιδανικό κόσμο και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι προτάσεις τις οποίες έχουμε μπροστά μας, οι προτάσεις της κυρίας Βέμπερ, μας δίνουν μια καλή βάση συζήτησης θα έλεγα με το Συμβούλιο έτσι ώστε να μην αγνοήσουμε την πραγματικότητα. Όταν πράγματι διαπιστούνται ένα σημαντικότατος κίνδυνος και όταν νιώθουν ότι απειλείται η ασφάλειά τους στα κράτη-μέλη, πρέπει να μπορούν να αντιδράσουν με τον σωστό τρόπο. Για τις λεπτομέρειες θα επανέλθουμε σε άλλη φάση. Πρέπει πρώτα όμως να συμφωνήσουμε, να καταλήξουμε σε ένα μηχανισμό ο οποίος στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνουμε μια πολύ σημαντική κατάσταση, ένα συμβάν το οποίο να θέτει σε απειλή την ασφάλεια μιας χώρας, να επαναφέρει η χώρα αυτή τους ελέγχους τους εσωτερικούς για να καλύψει αυτά τα κενά ασφαλείας τα οποία διαπιστώθηκαν. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι εντάξει δεν χρειάζεται συζήτηση. Όλα έχουν ε, ρυθμιστεί και μια μεγαλύτερη παρεμβατικότητα θα έλεγα από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα μπορούσε να αφαιρέσει κάποια δικαιώματα των κρατών μελών αυτό θα ήταν λάθος. Αντίθετα η πρόταση της κυρίας Βέμπερ προτείνει λύσεις αποδεκτές για όλους. έτσι ώστε να μπορέσουμε να δράσουμε όπως είπα ταχύτατα σεβόμενοι όλα τα προβλήματα ασφαλείας τα οποία μπορεί να δημιουργηθούν. Λοιπόν, ο τελευταίος ομιλητής πριν από την κυρία Βέμπερ. you go first, Mr. Mm. Silstra, would you like to comment? <coughs> Yes, I would. Thank you. Uh, Ο κύριο Ζήλστρα. Κύριε Πρόεδρε. Ναι, έχω μια περίεργη αίσθηση από τη συζήτηση αυτή που διεξιάγεται εδώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή είναι σαν να βρίσκονται από την μια μεριά και τα κράτη-μέλη από την άλλη μεριά. Αυτό δεν βοηθάει βέβαια καθόλου την Ευρώπη όπως καταλαβαίνετε. Η ασφάλεια είναι πολύ βασικό θέμα και είναι θέμα της ε, κυβέρνησης των χωρών. Την ασφάλεια την ε, προσφέρουν ε, τα κοινοβούλια και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Αυτό το οποίο μπορεί να καθορίσει, να καθοριστεί από τις Βρυξέλλες δεν μπορεί να είναι αυτό. Νομίζω ότι έτσι παρεμβαίνουμε στα δικαιώματα των κρατών μελών. Η επιθυμία των πολιτών, μα και τα δικαιώματα των πολιτών, είναι να μπορούν να είναι προστατευμένοι από κάποια δεχόμενη επίθεση. Δεν νομίζω λοιπόν ότι είναι καλή ιδέα τα θέματα της εθνικής ασφάλειας να περνάνε στις ε, Βρυξέλλες. Η μετανάστευση είναι άλλο θέμα, λαμπεντούσε κτλ αναφερθήκαμε στις αθλητικές διοργανώσεις. Μπορεί αυτό να είναι απειλή για τη δημόσια τάξη. Μπορεί μερικές φορές στην περίπτωση των χούλιγκανς και τα λοιπά, αλλά τότε είναι οι χώρες μέλη που πρέπει να το αναλάβουν. Μου φαίνεται πολύ περίεργη βάση πάνω στην οποία ετοιμάζεται η πρόταση αυτή. Δεν είναι δυνατόν οι Βρυξέλλες να αποφασίζουν πότε και για πόσο το κράτος μέλος θα αποφασίσει για την επαναφορά των εσωτερικών συνόρων. Δεν είναι δυνατόν να το κάνει, γιατί στο κάτω-κάτω ε, για το Σέγγεν έχουν να κάνουν και άλλες χώρες. Εγώ θα υποβάλω έτσι καλλιώς τροπολογία πάντως ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα κύριος Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι ξεκάθαρο από τη συζήτηση αυτή ότι υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων ότι το Σέγγεν πρέπει να διατηρηθεί. Ότι η ελεύθερη κυκλοφορία μπορεί να πάυσει μόνο σε ιδιαίτερα έκτακτες περιστάσεις και αυτό που είναι νέο είναι ότι όλοι συμφωνούμε για το ότι οι μεταναστευτικές ροές δεν μπορούν να αποτελέσουν αιτία για την επαναφορά των συνόρων στα εσωτερικά σύνορα. Και αυτό θέλω να ρωτήσω το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο παρακαλώ μπορεί να μας πει κατά πόσο την ίδια αίσθηση έχει και το Συμβούλιο για το θέμα αυτό της μετανάστευσης. Ποια είναι η άποψη των χωρών μελών όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι και η καρδιά του ζητήματος και θα ήταν καλό να μας το διευκρινίσει αυτό το Συμβούλιο. Έχοντας ακούσει τη συζήτηση, νομίζω ότι σε περίπτωση που η Προεδρία, η Επιτροπή θέλουν να σχολιάσουν, να το κάνουν πάρα πολύ σύντομα για να τηρήσουμε το χρόνο μας. Ε. Πολύ γρήγορα για τις ενστάσεις που ακούσαμε από αρκετούς εδώ όσον αφορά την ε, αιτιολόγηση της πρωτοβουλίας που ανελήφθη, τη λογική πίσω από την πρωτοβουλία αυτή, τα θετικά. Αν θέλουν, πριν επιστρέψουμε στην κυρία Βέμπερ, η Επιτροπή, η Προεδρία, ποιος, η Επιτροπή. Ναι, ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, θα απαντήσω σε κάποια ζητήματα και στα υπόλοιπα φαντάζομαι η Προεδρία θα το κάνει. Νομίζω λοιπόν ότι ορισμένοι ευρωβουλευτές δίνουν μια στραβή εντύπωση ε, του λόγου για τον οποίο προτίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το πακέτο αν ήταν απλώς και μόνο να αντιμετωπίσουμε μία ε, παράβαση που έγινε, δεν θα ήταν η σωστή βέβαια αντιμετώπιση. Θα ήθελα λοιπόν να ξαναδούν οι εξώτιμοι ευρωβουλευτές την ανακοίνωση για το πακέτο και από εκεί και πέρα διμερώς ευχαριστώ να συζητήσουμε μαζί τους για να εξηγήσουμε τους λόγους για τους οποίους οδηγηθήκαμε στην πρόταση αυτή. Νομίζω ότι η αντίδρασή τους είναι δυσανάλογη. Δεν πρόκειται για ένα-δύο επεισόδια. Είπαμε ότι δεν ε, ε, πρόκειται για καταστάσεις επαναφοράς των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Το Συμβούλιο τώρα. Ένα σύντομο σχόλιο παρακαλώ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Για την ερώτηση της κυρίας Μάκιντάις. Για το αν είναι ρεαλιστικό να καταλήξουμε σε συμβιβασμό και ότι κατά πόσο το σχέδιο είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Μα ακριβώ αυτό θα είναι και το αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Για τον κύριο Μπουσέτελ θέλω να πω ότι δεν υπάρχει στήριξη στο Συμβούλιο προκειμένου η μετανάστευση ως τέτοια να αποτελέσει αιτία για επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Η κυρία Βέμπερ τώρα, παρακαλώ. Ξέρω ότι δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους οι οποίοι τους τελευταίους μήνες πριν από την προετοιμασία της, αυτής της έκθεσης συνεργάστηκαν μαζί μου. Είχαμε πάρα πολλές συναντήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε πολλά επίπεδα. Επανειλημμένα συναντήθηκα και με την Προεδρία, με τους σκιώδεις εισηγητές επίσης από τις πολιτικές ομάδες. Τους ευχαριστώ όλους λοιπόν για την καθημερινή τους δουλειά και είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσουμε τη συνεργασία αυτή και στο μέλλον. Στην ουσία ακούστηκαν δύο απόψεις. Η πρώτη είναι αυτή η οποία λέγει ότι θέλουμε εμείς να ξεπεράσουμε αυτά τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα και θέλουμε να περάσουμε σε ένα συντονισμένο τρόπο αντίδραση στην περίπτωση επανεισαγωγής ελέγχων. Και η άλλη άποψη λέει ότι δεν χρειαζόμαστε αυτές τις ρυθμίσεις στην ισχύουσα κατάσταση. Αυτά τα οποία έχουμε είναι αρκετά και αυτά συνιστούν θα έλεγα την κατάσταση ως έχει και στα πλαίσια περιπτώσεων όπως αυτή της Λαμπεντούζα. Ας ασχοληθώ πρώτα με την δεύτερη άποψη. Είναι αλήθεια ότι εν μέρη αυτά τα οποία συνέβησαν ήταν απάντηση σε αυτά τα οποία συνέβησαν στη Λαμπεντούσα. Εγώ αναφέρθηκα σε αρκετά θέματα, σε αρκετά συμβάντα τον τελευταίο καιρό. Η επανεισαγωγή των ελέγχων στη Δανία δεν είχε καμία σχέση με τη Λαμπεντούσα. Ήταν μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης τότε να επανεισάγει τους ελέγχους αυτούς για την καταπολέμηση των εγκληματικών ενεργειών. Και όλοι συμφωνήσαμε ότι δεν ήταν σωστή η στάση αυτή. Αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει η έκθεση είναι να αποτρέψει την επανάληψη τέτοιων καταστάσεων στο μέλλον εμπλέκοντας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων και τα κράτη-μέλη. Όταν κάποια κράτη αποφασίσουν ότι θέλουν πράγματι να επανισάγουν τους εσωτερικούς ελέγχους. Κάποια πολύ συγκεκριμένα άλλα θέματα στα οποία δεν θα εξοδέψουμε πάρα πολύ χρόνο. Θα έχουμε το χρόνο να συναντηθούμε στο μέλλον για τη μη χρήση της επιτροπολογίας, κατανοώ τις απόψεις που ακούστηκαν, θα πρέπει να τις συζητήσουμε ε, περισσότερο. Νομίζω ότι κάτω από ιδιαίτερα έκτακτες συνθήκες ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να αναλάβει δράση. Θα δούμε πώς μπορούμε τη διαδικασία αυτή να την καταστήσουμε διαφανέστερη, αλλά πάντως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παραμείνει κύριος της διαδικασίας. Τώρα ε, δεν μιλάμε για κατεπήγοντα θέματα, δεν μιλάμε για τρομοκρατικές επι, επιθέσεις. Το δεκαήμερο ε, εσωτερικών επαναφοράς ελέγχων πολλοί πιστεύουν ότι είναι πολλές μέρες. Μαζί με κάποιες ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις στην Ισπανία Νομίζω ότι κάποιες τέτοιες τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ισπανία δεν ε, βοηθούνται σε τίποτα στην εξυχνίασή τους, δεν βοηθιέται σε τίποτα στην εξυχνίασή τους η επαναφορά για λίγες μέρες κάποιων εσωτερικών ελέγχων. Προφανώς τρεις μέρες είναι πολύ λίγο. Για την κυρία Μάκενταιρ στα πλαίσια της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρομαι στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ζητήσει την επανεισαγωγή ελέγχων. Αυτό είναι κάτι το οποίο το Συμβούλιο δεν δέχεται. Και όταν μιλάω για συντονισμένη αντίδραση, θεωρώ ότι το κράτος μέλος πρέπει να έχει πάντα την αρμοδιότητα να πάρει την απόφαση, αλλά μπορεί να το κάνει αυτό όταν η ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή επηρεάζεται άμεσα από την επανεισαγωγή των ελέγχων και εμπλέκεται συνεπώς. Τώρα για τις κατευθυντήριες γραμμές. Η ιδέα των κατευθυντηρίων γραμμών ε, δεν υπάρχει δεν την πήρα την ιδέα αυτή μέσω επιφύτησης. Υπήρχε στην ανακοίνωση της Επιτροπής. Αυτή ήταν η πηγή. Πέραν τούτου βέβαια κατανοώ ότι δεν θέλουμε να προχωρήσουμε ε, τόσο έτσι ώστε να ε, θεωρήσουν οι χώρες μέλη ότι απειλούνται οι αρμοδιότητές τους. Αλλά όταν μιλάμε για το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το και εκτιμένο Σέγγεν. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε παράλληλα ότι αυτό το οποίο συνιστά μία απειλή για μία δημόσια πολιτική ή για την εθνική ασφάλεια μίας χώρας είναι κάτι το οποίο επηρεάζει υποχρεωτικά το σύνολο της ζώνης Σέγγεν. Συνεπώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να κάνει μία προσπάθεια έτσι ώστε να προχωρήσει στη σύνταξη και πρόταση κατευθυντηρίων γραμμών. Γιατί αλλιώς η πρόταση την οποία κάνω αναφέρεται ε, συστηματικά σε απειλές σε κοινοτικό επίπεδο. Εφόσον υπάρχουν απειλές σε κοινοτικό επίπεδο πρέπει να υπάρξουν και κριτήρια για τον ορισμό αυτών των απειλών. Απλά λοιπόν δεν θα μακρηγορήσω. Θέλω να ευχαριστήσω τους γραμματείς μου και τους συμβούλους μου σε θέματα πολιτικής οι οποίοι ξενύχτησαν για να γίνει η πρόταση αυτή. Είχαμε μια συζήτηση πάρα πολύ χρήσιμη, υπήρξαν αντιτιθέμενες απόψεις, θα συνεχιστεί η συζήτηση, τώρα έχει ξεκινήσει. Έχοντας ακούσει λοιπόν ε, και τις απόψεις των κρατών μελών, η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών θα πρέπει να καθοριστεί η 12η μεσημβρινή της 9ης Μαρτίου. Η εξέταση των τροπολογιών θα πρέπει να γίνει στην επόμενη συνάντηση της Επιτροπής μας τα μέσα του μηνός Μαρτίου. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο με πέντε 5 λεπτά καθυστέρησης που θα πρέπει να καλύψουμε στην συζήτηση τι εκθέσεω του συναδέλφου κυρία Χολμάιερ για τι επιθεσει κατα κατά Σημάτων πληροφορικής 2005-222. Θα ακούσουμε την κυρία Χολμάιερ. Θα θυμάστε ότι η συζήτηση στόχο είχε όταν προβλέφθηκε να δούμε τις τροπολογίες. Ψηφοφορία δεν θα γίνει, μόνο ανταλλαγή απόψεων. Έχετε το λόγο κυρία Χόλμαϊερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ μαζί με τους κοιότητες συγκητές την προηγούμενη εβδομάδα ε, συμφωνήσαμε και δεδομένων των διαφόρων δεσμεύσεων ε, και κολλημάτων των συναδέλφων ότι θα πρέπει η ψηφοφορία να αναβληθεί. Μια και δεν είχαμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε με την ησυχία μας τις συμβαστικές τροπολογίες. Αυτό δεν, έχει, δεν αποτελεί ένδειξη ότι ε, ήμασταν διαιρεμένοι στις θέσεις μας, απλώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το χρόνο δεδομένου ότι ε, μεσολαβούσε μια πράσινη εβδομάδα. Και θα ήθελα ε, να προχωρήσω λέγοντας ότι ευχαριστώ και το Συμβούλιο για την κατανόηση που δείχνει, επισημένοντας βεβαίως Προ ε, του εκπροσώπους Συμβουλίου πως έχουμε αποφασίσει ότι μόνο δύο συνεδριάσεις τριμερούς διαλόγου θα χρειαστούν και θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε με το Συμβούλιο γιατί μπορούμε να είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και οδησηγητές για την συμμετοχή τους, για την αποφασιστικότητα και τη στράτευση με την οποία χειρίζονται το θέμα για το πολύ καλό πνεύμα που έχουμε μεταξύ μας και θα ήθελα να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι έχουμε να κάνουμε με ποινικό δίκαιο, δηλαδή εκείνο το, το μέσον επέμβαση, το οποίο αποτελεί σε τελευταία ανάλυση το τελευταίο βήμα. Εμείς βεβαίω θα προτιμούσαμε την ε, οδηγία πρόληψης και τις οδηγίες ε, για την ασφάλεια να, είχαμε, να συζητήσουμε ε, πριν να φτάσουμε στο ποινικό δίκαιο, αλλά τι να κάνουμε, οι ποινικέ ε, πτυχές μας έρχονται στην διαδικασία αυτή πρώτες και μετά θα πρέπει δυστυχώς να δούμε τις προτάσεις για την πρόληψη και αποτροπή. Θα τα δούμε και αυτά με τη σειρά τους. Εδώ έχουμε λοιπόν όπως είπα να μια οδηγία του ποινικού δικαίου. Το βλέπουμε άλλωστε και σε, ορισμένα αιτιολογικέ ε, σε ορισμένες αιτιολογικές αναφορές. Και ε, θα πρέπει οπωσδήποτε το κείμενο να διαμορφωθεί κατά τρόπο ασφαλή, σαφή, ε, δικαιικά για να μην υπάρχουν περιθώρια αμφισβήτησης ή παρερμηνίας. Κάποια ερωτηματικά που με απασχολούν θα ήθελα να φέρω, κάποιες τροπολογίες των συναδέλφων Βερζόν και Άλμπρεχτ συγκεκριμένα, που ζητούν την εξολοκλήρου απαλλαγή από ποινική ευθύνη κάποιου ο οποίος εγκαίρος και αυθορμήτως ενημερώνει τις αρχές για πιθανότητες ε, επίθεση στα συστήματά τους κτλ. Νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον ανεπαρκές ως πρόταση. Σε τελευταία ανάλυση μπορεί ένας επιτιθέμενος hacker το ΣΥΠΗΝ να ενημερώνει προ, πριν από την έναρξη της επίθεση του στι αρχέ, αλλά αυτό χωρίς βεβαίω να σημαίνει ότι επιδενώνεται η κατάστασή του, πάντω δεν τον απαλλάσσει και από κάθε ευθύνη. Μπορούμε να το δούμε όμως σαν ε, λόγους μείωσης της ποινής. Γιατί όντως υπάρχουν λόγοι μείωση τη ποινή που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και άρα καλό θα ήταν να μείνουν και αυτή, να μείνει αυτή η διάσταση, δηλαδή οι λόγοι μείωση τη ποινή, αλλά και οι επιβαρυντικέ συνθήκε. Εκείνε δηλαδή που θα οδηγούν σε πιο βαριά ποινή. Εν προκειμένου στην οδηγία δεν δημιουργούμε κανένα νέο ε, μόρφωμα, δεν εφευρίσκουμε τίποτα το καινούργιο δηλαδή. Ευχαριστώ για τις ε, παραπομπές ε, σε Europol και γενικά τις προτάσεις για δικτύωση, προ έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών, συνεργασία μεταξύ των αρχών, γιατί βέβαια στο δυνατόν πιο γρήγορο, στο δυνατόν με περισσότερη ακρίβεια και ευστοχία θα πρέπει να γίνεται η συνεργασία στο με αυτών. Μην ξεχνάμε ότι και εκείνοι οι οποίοι ε, αναπτύσσουν τι επιθέσει κατά των συστημάτων πληροφορική έχουν ε, σαν μεγάλο πλεονέκτημα και όπλο την καλή του δικτύωση, πολλέ φορέ είναι καλύτερη και από τη δική μα. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που θα πρέπει να συζητήσουμε. Άνσο και Άλβαρο με μια τροπολογία παραδείγματι που προτείνει να εφαρμόζεται η οδηγία αυτή και σε κρατικές τάξεις εφόσον είτε προξενούν είτε χρηματοδοτούν κράτη τέτοιου είδους επιθέσεις. Μακάρι, τι να σα πω, αν μπορέσουμε να το καταφέρουμε, αλλά μόνο στο πλαίσιο του Διεθνού δικαίου. Άλλη λύση δεν βλέπω. Ποινική δίωξη βάρο κράτου δεν προβλέπεται από ό,τι γνωρίζω μέχρι στιγμή στο διεθνέ δημόσιο δίκαιο. Το μόνο, η μόνη εξαίρεση που γνωρίζει το δίκαιο είναι αυτή του, των εγκλημάτων πολέμου, ε, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, για, για τα οποία έχει θεσπιστεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης. Δεν νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να στραφούμε ποινικά κατά μιας κρατικής τάξη μόνο, κατά ατόμων ιδιωτών δηλαδή και ανάλογα με τις δικαιοδοτικές ε, δυνατότητες με την έννοια ότι δεν, μπορούμε, δεν μπορεί ένα κράτος να θεωρήσει ως ε, ποινικά υπόλογο ένα άλλο κράτος και ότι ίσως συγκινησιακά να μα ενδιέφερε κάτι τέτοιο δυνατότητα τέτοια δεν υπάρχει. Επίσης, προσπαθώ να διευκρινίσω ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τη δυνατότητα άσκησης δίωξης κατά των επιμέρους αρχών διαχείρισης προσωπικών δεδομένων ή των ε, υπαλλήλων διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Εάν, ας πούμε, μια κρατική αρχή θέλει να αναπτύξει ένα σύστημα προστασίας προσωπικών δεδομένων και με στόχο να διαφυλάξει ολόκληρο το κρατικό σύστημα, όλες, όλες τις υπηρεσίες, ε, προτείνεται την, η ανάληψη του έργου από κάποιον ειδικό και Φερρυπίν προτείνεται τιμή 100.000 ευρώ που φαίνεται υπερβολική ε, σε μία αρχή δημοσιονομική, οικονομική, Υπουργείο Οικονομικών ότι είναι, το οποίο όμως τελικά λέει όχι είναι πολύ ακριβό, δεν μπορούμε να, χρηματοδοτήσουμε αυτό το έργο και άρα απορρίπτει την πρόταση. Τότε δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να ασκήσει δίωξη κατά του εν λόγω Υπουργείου ή της Υπηρεσίας ε, Προστασίας των Δεδομένων. Ο κύριος Άλμπρεχτ προκειμένου προτείνει μια καλή συμβαστική λύση νομίζω, ε, την οποία θα μπορούσαμε στην συγκεκριμένη αυτή υπόθεση να δεχθούμε. Κάποια επιμέρους ζητήματα ε, ασάφιες μπορέσαμε να διευκρινίσουμε ελάχιστη μέγιστη ποινή που σημαίνει ότι θα ορίσουν τα κράτη-μέλη ως το πολύ ανώτατη, μάλλον κατελάχιστον ανώτατη ποινή την τάδε. Το, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επιβληθεί και ανώτερη ποινή από την ε, κάθε εθνική εσωτερική τάξη, αλλά θα ε, προσδιορίζεται από την οδηγία ότι τουλάχιστον θα επιβάλλεται η τάδε ποινή. Αυτό για να μπορούμε με την ίδια αυστηρότητα να αντιμετωπίσουμε ποινικές ε, τέτοιες εγκληματικές πράξεις. πρόθεση ή καλύτερα απόπειρα. Η πρόθεση ίδια δεν μπορεί να ε, στοιχειοθετήσει απόπειρα παρά μόνο εάν ήδη έχει ξεκινήσει η παρίσφρηση στα ε, στοιχεία και το υλικό των δεδομένων. Το να συλλέξει δηλαδή κανείς ε, υλικό χωρίς όμως να μπει μέσα σε ένα σύστημα δεν επαρκεί για να στοιχειοθετήσει απόπειρα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι να επειδή μάζεψε κάποια ονόματα και αριθμός λογαριασμών ε, τραπεζικών έχει την πρόθεση να ε, σφεδερίσει τα χρήματα, να διάσει λογαριασμούς και άρα στη τα απόπειρα. Όχι, πρέπει να έχει ξεκινήσει και η επίθεση η ίδια. Γιατί όταν μιλάμε για προστασία δεδομένων πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ αυστηροί. Α, πρέπει η επίθεση κατά του συστήματος να σημαίνει να συνοδεύεται και από εγκληματική πρόθεση, από πρόθεση δηλαδή διάπραξης εγκλήματος. Διότι διαφορετικά, δεδομένου ότι δεν έχουμε να κάνουμε με την προστασία προσωπικών δεδομένων, ο καθένα θα μπορούσε να ε, επεμβαίνει, να μπαίνει σε όλε αυτέ τι βάσει δεδομένων που συλλέγονται με τα στοιχεία όλων μα σε τελευταία ανάλυση και να τι διαφυλάσσει για οποιοδήποτε λόγο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να υπάρχει η εγκληματική πρόθεση. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Χόλμαϊερ και τώρα παρακαλώ την Επιτροπή, την κυρία Γιάννη Σπερκινέλα. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως είπε και η κυρία Χόλμαϊερ, είχαμε πολύ επικοδομητικό διάλογο μεταξύ μας για τις τροπολογίες. Συζητήσαμε διάφορα ζητήματα από αυτά που ανέφερε και τώρα η κυρία Χόλμαϊερ. Σας ευχαριστώ. Στηρίζουμε την προσέγγιση επί της αρχής. Τίθεται διάφορα ζητήματα και για το θέμα ασυλίας ε, του κράτους, ε, της ευθύνης. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Πρέπει όμως να σκεφτούμε προσεκτικά, να μην το δούμε το θέμα πολύ στενά, το θέμα της ποινικοποίηση ε, δηλαδή, ίσως να μην είναι αυτός ο καλύτερος τρόπος. Υπάρχει ένα ολόκληρο φάσμα ε, παραβιάσεων και εγκλημάτων στον κυβέρνο χώρο. Σας ευχαριστώ πάντως που διευκρινίσατε το θέμα των ε, κυρώσεων. Υπάρχουν πολλές, κυρώσεις όσο, ε, πολλές συγγνώμη, τροπολογίες όσον αφορά τις κυρώσεις. Ένα από τα πράγματα που θα θέλαμε εμείς εδώ να διευκρινίσουμε είναι όταν βλέπουμε τροπολογίες που λένε ε, διαγραφή των κυρώσεων ή των επιβαρυντικών ε, συνθήκων. Ορισμένες από αυτές συμπεριλαμβάνονται ήδη στο πλαίσιο του 2005. Να έχουμε λοιπόν υπόψη μας ότι ένα από τα επιχειρήματα για την αύξηση των κυρώσεων ήταν και είναι η πραγματικότητα ότι οι κυρώσεις δηλαδή τώρα είναι πάρα πολύ χαμηλές και ότι το εύρος και η ζημιά από τις ε, επιθέσεις στον κυβερνοχώρο είναι κάτι πολύ σημαντικό για τόσο χαμηλές κυρώσει. Ευχαριστούμε κύριε Γιάνσκι. Ε, εκ μέρους του Συμβουλίου, ο κύριος Λάσκοφλη που εκπροσωπεί την Προεδρία της Δανίας. Παρακαλώ. Εκ μέρους της Προεδρίας και του Συμβουλίου θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για την υπόθεση αυτή και θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι είμαστε έτοιμοι να προωθήσουμε τις διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό. Από πλευράς της Προεδρίας λοιπόν θέλουμε να προχωρήσει η διαδικασία αυτή αισθητά κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας. Αναβάλλεται βέβαια η ψηφοφορία, δεν θα γίνει σήμερα, οπότε καταλαβαίνετε ότι το χρονοδιάγραμμα γίνεται πολύ σφιχτό. Πιστεύω όμως ότι θα καταφέρουμε με την καλή συνεργασία που είχαμε μέχρι τώρα να συνεχίσουμε έτσι και να πετύχει ο στόχος μας. Τώρα, οι τροπολογίε που προτείνουν τα μέλη της Επιτροπής αυτής δεν έχουν ακόμα αξιολογηθεί από την ομάδα εργασίας στο Συμβούλιο. Υπάρχουν όμως κάποια θέματα τα οποία θα μπορούσαμε ήδη να αναφέρουμε. Και ένα από αυτά, το είπε και ο συνάδελφο από την Επιτροπή και από την ίδια την κυρία Χολμάγερ, και είναι το θέμα της ε, ασυλίας των χωρών. Είναι θέμα δόγματος του διεθνούς δικαίου που βασίζεται στις αρχές της ισότητας και κυριαρχίας των χωρών. Εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο δόγμα, το δικαστήριο μπορεί να μην μπορέσει να ακολουθήσει νομολογία. Πάντως, όσον αφορά την νομολογία αυτή για ένα άλλο κράτος, η ασυλία είναι απόλυτη. Η οδηγία αυτή που θέλει να προχωρήσει προϋποθέσεις για τα κράτη-μέλη ώστε να μπορούν να διευθούν ποινικά, πρέπει να σέβεται το δόγμα του διεθνούς δικαίου. Εάν όχι, τότε προβλέπουμε ότι θα έχουμε τεράστιες δυσκολίες προκειμένου τα κράτη στο Συμβούλιο να υποστηρίξουν την πρόταση αυτή. Ένα άλλο θέμα που επανέρχεται στις τροπολογίες έχει να κάνει με τις ελάχιστες προδιαγραφές ε, προστασίας των ε, ε, προσωπικών δεδομένων και τις βάσεις δεδομένων. Λαμβάνοντας υπόψη λοιπόν τη νομική βάση της πρότασης αυτής, στόχος και το εύρος για την Προεδρία είναι ότι δεν πρόκειται για το κατάλληλο μέσο προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα που έχουν να κάνουν με την ευθύνη των φορέων. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Συζήτηση λοιπόν τώρα. Ο κύριος Κίρκοπ πρώτα απ' όλα. Κύριε Πρόεδρε, πέρα από τη δικιά μου έκθεση για τα δεδομένα PNR, αυτό είναι ένα επίσης πάρα πολύ τεχνικό θέμα που εξετάζουμε αυτή την εποχή. Βασιζόμαστε στο 2005 και την τότε σύμβαση. Αυτό είναι αναγκαίο γιατί τα εγκλήματα στον κυβερνοχώρο, όπως και η τεχνολογία, είναι πράγματα τα οποία προχωρούν με πολύ ε, ταχύς ρυθμούς. Μπορεί να πρέπει συχνά να ξαναβλέπουμε τις αποφάσεις μας αυτές, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα. Σίγουρα πάει προς τη σωστή κατεύθυνση η συγκήτρια. Πάντως θέλω να σχολιάσω δύο-τρία πραγματάκια. Πρώτον, ο λόγος που τα κάνουμε όλα αυτά είναι ότι την ευθύνη την μοιράζονται πολύ και διάφοροι οργανώσεις, άνθρωποι κτλ. Πριν από μία εβδομάδα πήγα στην Ευρωπαϊκή Έδρα της Intel, οι οποίοι φτιάχνουν μικροτσίπς, όπως ξέρετε. Και όλοι λένε ότι έχουν σχέσεις με επιχειρήσεις όπως είναι η Μάκαφη, που είναι επιχειρήσεις που δίνουν λογισμικό που βοηθάει να αποφεύγουμε ε, επιθέσεις ή ε, ναι, επιθέσεις σε διάφορα συστήματα πληροφορικής. Ξεκινάνε όλα από τους σχεδιαστές των ε, ηλεκτρονικών υπολογιστών και από τους ανθρώπους που ετοιμάζουν το λογισμικό. Είναι σημαντικό όμως να το ξέρουμε, γιατί το κυβερνοέγκλημα δεν μπορεί να λάβει χώρα αν όλοι κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να το σταματήσουμε. Και αυτό το οποίο είναι απογοητευτικό, και εγώ την πιστεύω την Intel, αυτό που είναι απογοητευτικό λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει αρκετή προσοχή από πλευράς των επιχειρήσεων μικρών και μεγάλων στην Ευρώπη αλλά και αλλού. Δηλαδή καθημερινά υπάρχουν χιλιάδες και δεν υπερβάλλω χιλιάδες επιθέσεις στον κυβέρνοχώρο στις βάσεις δεδομένων που έχουν αμερικανικά Ινστιτούτα και ευρωπαϊκά. Είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Παλιότερα όταν δύο κατάσκοποι συναντιόντουσαν σε μια γέφυρα και ο ένας έδινε στον άλλον έναν φάκελο σχετικά με το σχεδιασμό ενός μαχητικού αεροπλάνου. Πάει σε αυτός ο καιρός. Τώρα πατιούνται μερικά κουμπιά από ένα-δυο ανθρώπους οι οποίοι είναι αναμειγμένοι σε ένα εγκληματικό δίκτυο και τελείως έχουν στη διάθεσή τους μέσα σε χιλιοστά δευτερολέπτου ένα σωρό πληροφορίε. Πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε από τις επιχειρήσεις να κάνουν περισσότερα, να ξοδέψουν περισσότερα χρήματα και να ορίζουν κάποιον. Όλοι έχουμε αξιωματούχους που ασχολούνται με το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο, θα πρέπει να έχουμε σε όλε τι επιχειρήσει και κάποιον ο οποίο ασχολείται με τα συστήματα που χρησιμοποιούν για να αποφεύγονται τέτοιε επιθέσει στον κυβερνοχώρο. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι για το διεθνέ επίπεδο. Ωραία, καλά κάνουμε που έχουμε κάποιε κυρώσει, αλλά νομίζω ότι πραγματικά είναι πολύ χαμηλέ για νεόδορες σε σχέση με τα όσα συμβαίνουν όταν δισεκατομμύρια ευρώ διακυβεύονται. Είναι διεθνή η διάσταση αυτού του προβλήματο, βέβαια. Ξέρουμε ότι πολλές χώρες στον κόσμο βάζουν χρήματα ε, για το κυβέρνο έγκλημα και πρόκειται για έγκλημα, είτε το κάνει ένα άτομο, είτε το κάνει μια επιχείρηση, είτε το κάνει μια χώρα, είναι ένα έγκλημα. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν διεθνείς κυρώσεις που να εφαρμόζονται πιο πολύ από ό,τι μέχρι τώρα και όχι κάποιοι δικηγόροι μόνο να προσπαθούν να πάνε σε διεθνή δικαστήρια, γιατί αυτό είναι δύσκολο. Άρα λοιπόν τέτοιου είδους κλοπές ή τέτοιου είδους δράσεις που γίνονται με επιθέσεις στον κυβερνοχώρο είναι κάτι απαράδεκτο. Έπειτα υπάρχει και τρομοκρατία στον κυβερνοχώρο. Ορισμένοι θεωρούν ότι η τρομοκρατία είναι μια έκρηξη μετά από την οποία σκοτώνονται άνθρωποι. Δεν είναι μόνο αυτό όμω. Εγώ πιστεύω ότι η τρομοκρατία μέσω του κυβερνοχώρου είναι ένας τρόπος να υπονομεύονται θεσμοί, επιχειρήσεις, κράτη και αποτελεί εξίσου μεγάλο κίνδυνο, τον οποίο πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θα κατα... μπορούσε να καταστρέψει την εσωτερική μας αγορά, θα μπορούσε να καταστρέψει τη φύση της κοινωνίας μας. Και νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι ζωτική σημασία. Οπότε χαίρομαι για την πρωτοβουλία αυτή. Πιστεύω ότι είναι ένα σημείο κίνησης για μια διαδικασία η οποία θα μας οδηγήσει σε περισσότερη προσοχή. Και πιστεύουμε την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ευχαριστούμε κύριε Κύρκοφ, κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ. Και τον εισηγητή για την στενή συνεργασία. Νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά και έχουμε προχωρήσει και με ικανοποιητικό τρόπο. Θα ήθελα να επανέλθω σε αυτά τα οποία είπε ο κ. Σκέρκοπ για τις ευθύνες των επιχειρήσεων. Από την άποψη του Κοινοβουλίου η συζήτηση αυτή έχει γίνει επανειλημμένα ότι η οδηγία αυτή δεν θα πρέπει να περιορίζεται στον τομέα του ποινικού δικαίου και δεν θα πρέπει απλά να περιορίζεται στον καθορισμό ποινών. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο και για την πρόληψη. Πρέπει να δούμε και τι ευθύνε υπάρχουν από πλευρά αυτών που είναι υπεύθυνοι ε, για τη λειτουργία των συστημάτων έτσι ώστε να χρησιμοποιούν τις ε, τελευταίες διαθέσιμες τεχνολογίες λοιπά. Να μην περιοριζόμαστε λοιπόν στον τομέα τον ποινικό. Γιατί τελικά θα αντιμετωπίσουμε προβλήματα σε σχέση με την εξέβρεση της σωστής λύσης. Το ποινικό δίκαιο δυστυχώς Ποτέ δεν λύνει πραγματικά το πρόβλημα. Το ποινικό δίκαιο στην ουσία επιβάλλει κάποιες ποινές αλλά δεν λύνει τα προβλήματα στη γένεσή τους. Πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε εμείς να βελτιώσουμε εκ των προτέρων την κατάσταση, να διαβρύνουμε το εύρος ακριβώς το μέγεθος της πρότασης αν θέλετε, το πεδίο καλύτερα της πρότασης, γιατί η επιβολή ανώτερων κάθε φορά ποινών από μόνη της δεν είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει ιδιαίτερα. Δεν είμαι βέβαιος ότι σαν παράδειγμα στην περίπτωση των επιβαρυντικών συνθήκων δεν νομίζω ότι είναι ένα κριτήριο το οποίο μπορούμε να εφαρμόσουμε στην περίπτωση της μη αποκάλυψης της ταυτότητας αυτών οι οποίοι κάνουν παράνομου τύπου προσβάσεις σε αρχεία ή σε ε, τράπεζες δεδομένων κτλ. Δεν είναι λοιπόν σωστός ο τρόπος αυτός από μόνος του. Θα πρέπει να υπάρξει μια διαφοροποιούμενη αντιμετώπιση των περιπτώσεων ε, στις οποίες υπάρχει μια παράνομη επίθεση αν θέλετε με πρόθεση την πρόκληση ζημιών και να την ξεχωρίσουμε από την ίδια περίπτωση μεν αλλά χωρίς ε, πρόθεση πρόκληση ζημιών. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική αντιμετώπιση των δύο καταστάσεων γιατί αλλιώς θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Θυμίζω ότι και στο Αμερικανικό Κογκρέσο στη φάση αυτή υπάρχει μια προσπάθεια αντιμετώπισης των θεμάτων αυτών οι οποίοι δεν σκοπεύουν να προκαλέσουν πραγματική ζημία σε ε, μια τράπεζα δεδομένων, αλλά χρησιμοποιούν παρόλα αυτά χωρίς να δικαιούνται ένα σύστημα, ε, κάποιες ιστοσελίδες, χωρίς όμως την πρόθεση να προκαλέσουν ζημίες. Ευχαριστώ κύριο Σέλσιο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας για τις προσπάθειες τις οποίες έχει κάνει και για τον πολύ σωστό τρόπο με τον οποίο εργάστηκε μέχρι τώρα. Όπως ε, έχουμε πει μέχρι τώρα, θα ήθελα να προσθέσω και εγώ κάποια σχόλια, γύρω από τα οποία μάλιστα έχω ήδη καταθέσει και ορισμένε τροπολογίες. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες αρχές από τη μία για τα θέματα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο σε ευρωπαϊκό και σε εθνικό επίπεδο στα πλαίσια του Eurojust σαν παράδειγμα, όλες αυτές οι υπηρεσίες θα πρέπει να εμπλακούν και να συνεργαστούν. Δεν πρέπει να αγνοήσουμε επίσης ότι το φαινόμενο του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο είναι ένα συνολικό παγκόσμιο φαινόμενο. Απαιτείται συνεργασία λοιπόν σε διεθνές επίπεδο γιατί αλλιώς δεν θα πετύχουμε τίποτα. Παράλληλα έχουμε προτείνει όλες οι διεθνείς συμφωνίες τις οποίες προσυπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη που περιλαμβάνουν ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και ό,τι έχει σχέση με την διασφάλιση ακριβώς της σωστής λειτουργίας του διαδικτύου. Όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, Κάτι τέτοιο διαφεύγει αν θέλετε της εμβέλειας της οδηγίας, αλλά το θέμα της πρόληψης, γιατί περί αυτού πρόκειται, είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι ο ρόλος τον οποίο παίζει η ΕΝΙΣΑ θα πρέπει να ενισχυθεί. Η ΕΝΙΣΑ θα πρέπει να δημοσιεύει συνεχώς εκθέσεις για το τι ακριβώς συμβαίνει σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο. Και η τεχνική εμπειρογνωμοσύνη της ΕΝΙΣΑ θα πρέπει να γίνεται γνωστή και να μοιράζεται αν θέλετε στα κρατημένη. Ίσως δεν ήμουν αρκετά αναλυτικός στο παρελθόν για την πρόταση συμπερίληψης και της ευθύνης των κρατών, όχι μόνο των επιχειρήσεων. Υπάρχει η άποψη με την οποία συμφωνούν και άλλες πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Άλμπρεχτ έχει υποστηρίξει την πρόταση αυτή στην πρόταση την οποία είχα κάνει εγώ, είχα ζητήσει όχι να θεωρείται υπεύθυνο και υπόλογο ένας κράτος μέλος, ένα κράτος μέλος και να παραπέμπεται ε, σύμφωνα με το ποινικό δίκαιο. Θα ήθελα όμως να αναγνωρίσουμε ότι το κράτος εκπροσωπείται από κάποια θεσμικά όργανα και αυτά τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να είναι υποχρεωμένα να προστατεύσουν τα συστήματα τηλεπικοινωνιών και τα συστήματα πληροφορικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε ενδοκινοτικό και σε διεθνές επίπεδο. Υπάρχουν πολλά συστήματα λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα οποία χρησιμοποιούνται από όλα τα κράτη-μέλη και τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν αντικείμενο επίθεσης από το, από το εσωτερικό των κρατών μελών. Συνεπώς δεν μπορούμε να μιλάμε απλά για την ευθύνη των νομικών προσώπων. Προφανώς και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προστατεύουν τα συστήματα λειτουργία τους, αλλά και οι κρατικές υπηρεσίες και τα θεσμικά όργανα τα δημόσια θα πρέπει να είναι υπεύθυνα να αναγνωρίζεται γι' αυτά μια συγκεκριμένη ευθύνη στην περίπτωση κατά την οποία κληθούν να διαχειριστούν ένα σύστημα το οποίο δεν είναι αυστηρά εθνικό αλλά κοινοτικό. Τώρα για το επίπεδο των κυρώσεων, των προστήμων. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να υποστηριχθούν. Όμως όπως όλοι γνωρίζουμε οι ποινές και οι κυρώσεις από μόνες τους δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο. Οι συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες προτάθηκαν από την κυρία Χολμάγερ νομίζω ε, οδηγούν στη σωστή κατεύθυνση. Και νομίζω ότι στο τέλος θα έχουμε ένα ισόρροπο κείμενο, ένα κείμενο που θα αποτελεί τη σωστή βάση για διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Κυρία Ένωση, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Εκ μέρους κυρίας Βεζατή, σκιώδης συζητήτρες, θέλω να κάνω μερικές παρατηρήσεις. Καταρχάς βλέπουμε βεβαίως ε, και εμείς ε, τον κίνδυνο της, ε, του να, της κυβερνοεγκληματικότητας. Αλλά δεν νομίζουμε ότι μπορούμε να τον απαλείψουμε ή να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα μέσω μόνο του ποινικού δικαίου. Είναι μονομερής η στροφή προς το ποινικό δίκαιο και πρέπει να την αναθεωρήσουμε. Έχουμε επίσης ενδιασμούς προς το ύψος των ποινών και δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε την επιδιωκόμενη λύση. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε με πιο διαφοροποιημένο τρόπο την κατάσταση, να έχουμε μια πιο διαφοροποιημένη προσέγγιση και ιδιαίτερα, ιδιαίτερα να δώσουμε προσοχή στο ότι δεν θέλουμε να ποινικοποιηθεί ο χρήστης και ο πάροχος των υπηρεσιών. Υπάρχει κίνδυνος, τον βλέπουμε ορατό, εάν παραμένει το κείμενο όπως έχει, όπως έχει σχεδιαστεί μέχρι τώρα και γι' αυτό θα κοιτάξουμε πολύ μεγάλη προσοχή έτσι ώστε να βρούμε μία λύση όσο το δυνατόν ευρύτερη Και γι' αυτό θα ήθελα εκ μέρους της, Επιτροπή, της ομάδας μας να επισημάνω ότι θέλουμε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Α, την επόμενη εβδομάδα θα βρεθούν οι σκιώδεις συγκητές στην αναζήτηση, μια συνεδρίαση με στόχο την αναζήτηση συμβαστικών τροπολογιών. Θα θέλαμε περισσότερο χρόνο για να μπορέσουμε και σε επίπεδο της ομάδας μας να καταλήξουμε σε μια τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χολμάιερ. Πρόεδρε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επισημάνω ορισμένε παρατηρήσει και να απαντήσω σε κάποια από τα σχόλια των συναδέλφων. Ε, τα όσα είπα ο κύριο ε, Κέρκοπ και ο κύριο Έντσιου σε σχέση με το τι κάνουμε σε περίπτωση παραβίαση από ή επιθέσεων από κράτη. Δεν μπορεί να ενταχθεί μέσα σε μια τέτοια οδηγία του κοινού δικαίου αυτό το θέμα. Αλλά ίσως στο πλαίσιο των διεθνών διασκέψεων μπορούν τα κράτη, οι εκπροσωποί μας να φέρουν το θέμα αυτό, έτσι ώστε να ρυθμιστεί μέσα στο διεθνές δίκαιο. Έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν ανησυχίες ε, κρατών μελών που διαπιστώνουν ότι δεν είναι σε θέση να ε, ασκήσουν δίωξη εις βάρος άλλων κρατών σε περίπτωση επιθέσεων μέσω του ε, διαδικτύου. Αυτό νομίζω κατά των συστημάτων πληροφορικής. Αυτό είναι κάτι το οποίο ε, μπορούμε να διεκδικήσουμε μέσω του διεθνού δικαίου. Νομίζω ότι είναι σαφέ και για τον κύριο Κέρκοπ και για τον κύριο Έντσιο. Θα πρέπει η ρύθμιση να γίνει μέσω του διεθνού διακρατικού δηλαδή δικαίου. Στο ζήτημα της ε, κλοπής ταυτότητας, από ό,τι βλέπω, από αυτά πρέπει να και οι νομικοί ειδικοί, στο identity theft, κλοπή ταυτότητα. δεν εννοούμε το να χρησιμοποιήσει κανείς το password του ενό ή του άλλου ή ε, να προσλάβει ένα κωδικό όνομα το οποίο ενδεχομένω δίνει άλλα στοιχεία για την προσωπικότητά του. Δεν ε, αφορά τέτοιου είδου υποθέσει, άλλωστε αυτέ είναι αποκλεισμένε εξ αρχή από το κείμενο. Εδώ όμω έχουμε να κάνουμε το cloud και με διάφορε ε, ρυθμίσεις που θα αντιμετωπίζουν το φαινόμενο κάποιοι να μπορούν να μπουν σε υπολογιστές ηλεκτρονικούς και μάλιστα κατά εντατοντάδες με στόχο να κλέψουν ε, στοιχεία ε, οικονομικά, δεχομένως για σκοπούς μηχανικής κατασκοπίας και ούτω καθεξής. Ε, που πολλέ φορέ προξενούν μάλιστα και τεράστιε οικονομικέ ζημιές. Εδώ λοιπόν προφανώ ε, δεν ε, μπορούμε να έχουμε μια πολύ χαμηλή ποινή. Μάλλον θα είναι μάλιστα επιβαρυντικές οι συνθήκε τη κλοπή ή υποκλοπή προσωπικότητα. αλλά είναι κάτι που θα συστήσουμε με την Επιτροπή. Στη μονομερή ε, τοποθέτηση ως προς το ποινικό δίκαιο, την κυρία Ένστη και την παρατήρηση της, θα ήθελα να πω ότι για τις λοιπές οδηγίες μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι τις ετοιμάζει, είναι το θέμα δηλαδή της ασφάλειας της πρόληψης, θα μας υποβάλει τις σχετικές προτάσεις και μέχρι το τέλος του έτους πιστεύω θα έχει ολοκληρωθεί. Η ποινική διάσταση προκύπτει μετά τη διάσκεψη της Βουδαπέστης ως μια ανάγκη για συνέχιση των εντατικών συζητήσεων που θα αναπτυχθεί εκεί και ίσως δεν είναι τόσο ε, περίπλοκο θέμα όσο αυτό του cyber security της κυβερνοασφάλειας. Έχουμε μια κάποια εμπειρία συλλέξη και από τα κράτη-μέλη έχουμε μπορέσει, από ό,τι διαπιστώνουμε, να αποκλείσουμε κάποιες σχετικά ελαφρές περιπτώσεις ε, επιθέσεων. Δεν προσπαθούμε να ε, ποινικοποιήσουμε συλλήβδιν χρήστες και παρόχους. Με τους παρόχους θα μιλήσουμε και λίγο περισσότερο. Ενδεχομένως να χρειαστούν κάποιες χρηματικές ποινές σε πολύ συγκεκριμένε ε, περιπτώσεις. Για δε το χρήστη ένας κοινό χρήστης δεν θα έχει κίνδυνο να του επιβληθεί ποινική κύρωση. Αν μπαίνει στο ίντερνετ, συμπεριφέρεται κανονικά, δεν διαπράττει κανένα έγκλημα. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα, θα πρέπει την επόμενη εβδομάδα, και γι' αυτό ζητώ την κατανοή να είμαστε έτοιμοι για να προλάβουμε μέσα στο χρονικό περιθώριο που έχει η Προεδρία τη Δανία να ολοκληρώσουμε όλο αυτό το εγχείρημα, διότι τα κύρια ζητήματα νομίζω είναι ξεκάθαρα και έτσι μέσα στι επόμενε μία ή δύο εβδομάδε μπορεί το Κοινοβούλιο να έχει ολοκληρώσει τη δουλειά του, να γίνει ψηφοφορία μα εδώ για να μπορέσουμε μετά να ξεκινήσουμε τι πραγματεύσει με το Συμβούλιο. Χαίρομαι ιδιαίτερως για τη συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφου για την βοήθεια που προσέφεραν και ιδιαίτερα βέβαια τη γραμματεία μας, αλλά και το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς λέει ο Πρόεδρος, ολοκληρώνουμε έτσι και ακούσαμε τη συζήτηση. Ψηφοφορία δεν προβλεπόταν, ανταλλαγή απόψεων μόνο. Αντιλαμβανόμαστε ότι η εισηγήτρια θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε μαζί με τους σκιώδεις εισηγητές να έχει κλείσει το θέμα μέχρι τα τέλη Μαρτίου για να συνεχιστεί η συζήτηση και να είμαστε έτοιμοι σε μια προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών να κλείσουμε το θέμα. Και τώρα περνάμε στο σημείο που αναβλήθηκε από χτες και που μπήκε στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για το σημείο της συναδέλφου μας, της κυρίας Χάνκης. Πρόκειται για την προστασία υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας, επιτεύγματα και επόμενα βήματα προς την παγκόσμια ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Θα ακούσουμε την παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης και μετά Ξέροντας ότι η Ήτρα είναι η αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, εμείς γνωμοδότηση υποβάλλουμε, θα πρέπει να ορίσουμε προθεσμοί για την υποβολή τροπολογιών. Σας υπενθυμίζω ότι έχουμε καθυστερήσει λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει 12 και 30 ακριβώς πρέπει να ξεκινήσουμε τη συνεδρία των συντονιστών σήμερα, γιατί έχουμε πολλά θέματα εκεί. Οπότε για να μας δοθεί μία ώρα χρόνος για τους συντονιστές θα πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει μέσα στο 12.30. Άρα να βιαστούμε. Πρώτα απ' όλη η η κυρία Χάνκης έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Επιτροπή Ήτρε είναι αρμόδια επί της ουσίας Επιτροπή για να ετοιμάσει την έκθεσή της. Εμείς μόνο γνωμοδοτούμε και είμαστε υπεύθυνοι για τις ζωτική σημασίας υποδομές. Ε, ο κυβερνοχώρος είναι ένας από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωτερική ασφάλεια. Η νομοθεσία όσον αφορά τις επιθέσεις στο κυβερνοχώρο είναι ένα θέμα που εξετάζει η ΛΥΠΕ στα πλαίσια της ε, έκθεσης που ετοιμάζουμε για οδηγία από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο όσον αφορά την αντιμετώπιση επιθέσεων στα συστήματα ε, πληροφορικής με συγκίτρια την κυρία Χολμάγερ. Έχετε μπροστά σας την πρόταση γνωμοδότησης. Εδώ προσπαθώ να υπογραμμίσω την διαπιστημονική προσέγγιση όσον αφορά τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και όσον αφορά την ασφαλειά μας αυτών. Γιατί είναι ζωτική σημασία υποδομές πληροφοριών. Μεταξύ άλλων, έχει να κάνει το θέμα με την μεταφορά δεδομένων και την αποθήκευση δεδομένων. Πρόκειται συχνά για ευαίσθητα δεδομένα που έχουν να κάνουν είτε με τις κυβερνήσεις στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε με δημοσιονομικούς οργανισμούς. Άρα όλα αυτά αποτελούν μέρος της ζωτικής σημασίας υποδομών πληροφοριών. Σε καθημερινή βάση χειριζόμαστε τέτοια δεδομένα και πρόκειται πολλές φορές ε, όχι μόνο για πραγματικές υποδομές αλλά και για εικονικές ε, υποδομές. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς γίνεται η ροή των ε, πληροφοριών των δεδομένων αυτών, να δούμε πώς θα χρησιμοποιείται το σύννεφο, το clouding, για την αποθήκευση επίσης πληροφοριών και δεδομένων. Θέλουμε λοιπόν προστασία των υποδομών και των πληροφοριών, όχι μόνο γεωγραφικά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας και ότι θα υπάρχει καλός συντονισμός μεταξύ των στρατιωτικών και των μη στρατιωτικών φορέων, όπως επίσης ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Η συνεργασία και ο συντονισμός είναι κάτι που χρειάζεται πάρα πολύ για να αποφεύγονται επικαλύψεις και συγχρόνως να μην υπάρχει έλλειψη πληροφοριών. Πρέπει γι' αυτό να υπάρχει ένας αξιωματούχος ε, να διοριστεί δηλαδή αρμόδιο αξιωματούχο για τον συντονισμό, πιθανώ με καθήκοντα συντονισμού τη ασφάλεια του κυβερνοχώρου σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Τη γνωμοδότησή μου την έχετε ε, γραπτά μπροστά σα, φαντάζομαι, οπότε δεν χρειάζεται να μπω σε λεπτομέρειε. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you, Mrs. Now Ευχαριστούμε, κύριε Χανκή. Τώρα, ποιο θέλει να πάρει το λόγο. Η κυρία Ρομέρο βλέπω είναι η πρώτη. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι μια αναγκαία έκθεση τη σήμερον ημέρα, διότι οι υποδομές ζωτικής σημασίας, οι υποδομές πληροφοριών, όντως μπορεί να αποτελέσουν θύματα επιθέσεων στο κυβερνοχώρο. Εδώ βέβαια έχουμε να κάνουμε και με τα συμπεράσματα που βγάλαμε στην προηγούμενη έκθεση. Προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αποτελεί κατά προτεραιότητα στόχο ενός hacker η Ευρωπαϊκή Δημόσια Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε συστήματα προστασίας, επίγει μάλιστα. Η πρόταση λοιπόν που έγινε και το σχέδιο που ακολουθεί η οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το βλέπουμε και στις ανακοινώσεις της Επιτροπής Όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται ενίσχυση, γιατί κάποιες χώρες δεν έχουν καν ομάδες κέντρα που να ανταποκρίνονται σε αυτό το στόχο προστασία των υποδομών προφοριών ζωτική σημασία. Γι' αυτό και είναι αναγκαία η συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και συγχρόνω, όπω λέει και η έκθεση, πρέπει να προσπαθήσουμε η συνεργασία αυτή να έχει και μια συνολική διάσταση σφαιρική, γιατί οι επιθέσεις που γίνονται στο κυβερνοχώρο γίνονται σφαιρικά. Το να υπάρχει <clears throat> ένας αξιωματούχος αρμόδιος για το συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό και όπως λέει η έκθεση της κυρίας Χάνκης, είναι σημαντικό να υπάρχει και καλύτερο συντονισμός μεταξύ των στρατιωτικών και μη στρατιωτικών φορέων όσον αφορά την ε, ε, παροχή πληροφοριών και δεδομένων. Υπάρχουν κάποιες ζώνες, βλέπετε, που υπάρχουν τριβές. Γι' αυτό καλό είναι να υπάρχει συνεργασία μεταξύ όλων των φορέων στατιωτικών και μη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να υπάρχει το κριτήριο της διαεπιστημονικής προσέγγισης, όπως λέει η κυρία Χάκης, αλλά να υπάρχει και συντονισμός ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορεί να ε, δώσει μια απάντηση και να προσφέρει προστιθέμενη αξία σε όσα γίνονται σε ολόκληρο τον κόσμο όσον αφορά την προστασία των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας. Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η έκθεση αυτή και ελπίζω να μπορέσω να υποβάλω ε, κάποιες ενδιαφέρουσε ε, τροπολογίες, αν και η κυρία Χάκη είναι αλήθεια ότι έχει επικεντρωθεί πολύ καλά στο θέμα και έχει συμπεριλάβει τα πιο σημαντικά ζητήματα. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Άλλες παρεμβάσεις. Κανένας άλλος. Καλώς. Κύριε Χάνκης, εσείς θέλετε να σχολιάσετε πριν περάσουμε στο επόμενο σημείο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρομέρο, για τόσο μας είπατε. Να προσθέσω μια πρόταση μόνο, ειλικρινά. Φοβόμουν ότι η ιδέα μου αυτή για τον συντονιστή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα την απορρίπτατε. Γιατί ακόμα δεν ξέρω κατά πόσο είναι αποδεκτή μεταξύ μας. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ που η κυρία Ρομέρο Λόπες τη δέχεται και συμφωνεί με αυτήν. Περιμένω λοιπόν τροπολογίες και φαντάζομαι ότι θα καταλήξουμε σε κάποια συμβαστική τελικά πρόταση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε κυρία Χάνκης και πάλι δεν υπάρχουν άλλα σχόλια. Σας υπενθυμίζω μόνο ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών θα είναι 29 Φεβρουαρίου. Αύριο δηλαδή. Αύριο, Τετάρτη, 12 το μεσημέρι. 12 το μεσημέρι. Σύμφωνοι. Συμφωνείτε. Καλώς. Και περνάμε στο επόμενο σημείο, το σημείο 14. Ευχαριστούμε κυρία Χάνκης. Δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών και δικαίωμα επικοινωνίας μετά τη σύλληψη. Έχουμε ένα σχέδιο έκθεσης για πρόταση οδηγίας όσον αφορά το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο είναι το τρίτο βήμα προκειμένου να εφαρμόσουμε τον χάρτη πορείας. Πρόκειται για πρόταση του Συμβουλίου του 2009 και μετά την οδηγία για το δικαίωμα σε διερμηνία και μετάφραση στα δικαστήρια, πρόταση του 2010. Και υπάρχει και το δικαίωμα πληροφοριών σε σχέση με δικαστικές διαδικασίες. Υπάρχει δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα. Τώρα θα ακούσουμε την εισηγήτριά μας, την κυρία Αντωνέσκου. Και μετά θα ακούσουμε την Επιτροπή και την Προεδρία. Και συζήτηση βέβαια. Λοιπόν, κύριε Αντωνέσκου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε ένα σχέδιο οδηγίας, πρώτας οδηγίας, που στόχο έχει τον προσδορισμό ελάχιστων προδιαγραφών σχετικών με τα δικαιώματα των ε, κατηγορουμένων σε ποινικέ ε, υποθέσεις. Πρόκειται για το τρίτο μέτρο που εγγράφεται στον, ε, στο φιλοπορίας για τα ποινικά. Έχουμε κοινέ αρχές που απορρέουν από τον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Δικαιωμάτων, και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Τα δικαιώματα όμως που αναγνωρίζονται στους πολίτες διαφέρουν από κράτος σε κράτος, καθώς η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν τη χάνει του ίδιου σεβασμού από τα κράτη-μέλη. Η νομοθεσία που εγκρίνεται από την Ένωση, που εισάγεται από την Ένωση, βελτιώνει την ε, αποτελεσματικότητα και τον ε, και της ε, επιβολής των ποινών και της δίωξης, αλλά έχει πολλές φορές ε, επισημάνει το Κοινοβούλιο την ανάγκη να βελτιώνεται η προστασία των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου στις ποινικέ υποθέσεις, γιατί βλέπουμε μια ξεκάθαρη απουσία ε, ισο και γι' αυτό θα πρέπει να μιλούμε πρώτα για μια πιο ενιαία αντιμετώπιση και μετά για μέσα αναμοιβαίας αναγνώρισης. Έτσι λοιπόν θέλουμε να βελτιωθούν τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, λαμβανομένης υπόψη όμως και της ανάγκης για ορθή απονομή δικαιοσύνης και για προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Τα δικαιώματα του κατηγορουμένου, εάν δεν έχει πρόσβαση σε δικηγόρο, μετατρέπονται σε μια απλή φερνάκι. Και γι' αυτό θα πρέπει να εξασφαλιστεί πάνω απ' όλα το δικαίωμα πρόσβαση στη δικηγόρο. Και έτσι με τι τροπολογίε μου προσπαθώ να κάνω τα εξή. Καταρχά γιατί θέλω να διαφυλάξω τη συνέπεια με τα πρώτα μέτρα, δηλαδή την οδηγία ε, για το δικαίωμα σε μετάφραση και διερμηνία και το δικαίωμα για ενημέρωση του υπόπτου. Ε, όσο δε αφορά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, θεωρώ ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προσφέρουν ε, και να εγγυώνται ευρύτατα δικαιώματα για τον κατηγορούμενο. Ο κατηγορούμενος θα πρέπει να έχει άμεση πρόσβαση σε δικηγόρο πριν από την ε, ανάκρισή του από τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές. Όταν του απαγγέλλονται κατηγορίες για έγκλημα ή όταν αποφασίζεται η προσωρινή του κράτηση, και πάντως για κάθε επικοινωνία του με τις αρχές. Και ο κατηγορούμενος ή ύποπτος θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να προσέλθει στο δικαστήριο συνοδευόμενος από τον συνήγορό του. Έχουμε τις ε, τροπολογίες λοιπόν ε, μέχρι την 27 που στόχο έχουν ε, την εναρμόνιση με τις ιδέες αυτές 26-27 που αφορούν μικρότερης βαρύτητας αδικήματα και σε άλλες ε, χώρες προβλέπεται αρχή όχι ποινική ως αρμόδια για την επιβολή κυρώσεων για τα λιγότερο σημαντικά παραπτώματα διοικητικού χαρακτήρα κυρώσεις δηλαδή και γι' αυτό δεν απαιτείται, δεν, φρονούμε, δεν θεωρούμε απαραίτητο και λογικό να προβλέπεται συνήγορο σε κάθε τέτοια περίπτωση στα διοικητικά παραπτώματα, στα απλά παραπτώματα ή και πτέσματα. Επίσης, Όταν υπάρχει περίπτωση για κάποιο πτέσμα επιβολής κυρώσεως ποινικής και παραπομπή σε δικαστήριο, τότε ε, μετατρέπεται σε υποχρεωτική η και πτεσματα επισης οταν υπαρχει περιπτωση για καποιο πτεσμα επιβολης κυρωσεως ποινική και παραπομπη σε δικαστηριο τοτε ε μετατρεπεται σε υποχρεωτικη παρουσια του συνηγόρου. το δικαίωμα της εκπροσώπησης από δικηγόρο ε, στις ποινικέ υποθέσεις κατά τη διάρκεια της προδικασίας, διερεύνηση δηλαδή της υπόθεσης, πρώτη διερεύνηση αμέσως μετά την τέλεση της πράξης ή σε περίπτωση σύλληψης από αυτοφόρο, δεν μπορούν αυτές οι πράξεις να θεωρηθούν ως ανακριτικές και αυτά προσπαθώ να τα διευκρινίσω στην ε, τροπολογία 12, αιτιολογική σκέψη Γ, Σ. Η συνομιλία, δηλαδή υποβολή ερωτήσεων από τις διοκτικές και δικαστικές αρχές ε, αμέσως μετά τη διάπραξη της πράξης, δεν μπορούν να θεωρούνται ως ανάκριση. εφόσον αφορούν μόνο ζητήματα ασφαλείας για το εάν υπάρχει ε, ε, κατοχή όπλων νόμιμη ή μη ή αν πρόκειται για επαλήθευση ταυτότητας. Και εδώ συμφωνώ με σχόλια των συναδέλφων ε, που ε, λένε ότι θα ε, ε, σήμαινε σημαντικό φόρτο για τις αρχές των κρατών μελών το να απαιτηθεί για κάθε περίπτωση επαλήθευση ταυτότητας από τις αρχές στο δρόμο ενός οποιοδήποτε υπόπτου να είναι παρόν και ο δικηγόρος του. για τα αποδεικτικά στοιχεία και την παρουσία δικηγόρου στην συλλογή αποδεικτικών προκειμένου να αποφεύγονται καθυστερήσεις αλλά και αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση Φερρυπίν στην περίπτωση της συλλογής ε, της, ε, των δακτυλικών αποτυπωμάτων ή της, ε, του αλκοτέστ ελέγχου αλκοολομετρίας. Λέμε ότι θα χρειάζεται παρουσία δικηγόρου μεν, αλλά με τις τροπολογίες μου 14 και 31 επισημαίνω ότι μετά το διορισμό του ο δικηγόρος μπορεί να ζητήσει να ενημερωθεί για την ενέργεια των πράξεων αυτών και θα πρέπει να ενημερώνεται, να του κοινοποιείται δηλαδή η διεξαγωγή τέτοιων πράξεων από τις αρμόδιες αρχές. Αυτό μετά την, ε, τις συζητήσεις που είχαμε με τους σκιώδεις συγητές μπορούμε να το βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο επισημένοντας ότι η πράξη συλλογή των αποδεικτικών όταν δεν υπάρχει διορισμός ε, δικηγόρου προηγουμένως αποτελεί την πρώτη πράξη για την οποία πρέπει να ενημερωθεί ο δικηγόρος και ε, θα καταθέσει σχετική τροπολογία. Το δικαίωμα της επικοινωνίας με τον δικηγόρο μετά τη σύλληψη. Ε, μετατρέπεται σε δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου μετά τη σύλληψη για λόγους προσαρμογής στο κείμενο των λοιπόν τροπολογιών. Τροπολογία 33 και το άρθρο 4. ορίζει ότι ούτε η διάρκεια και η συχνότητα των διαβουλεύσεων μεταξύ υπόπτου ή κατηγορουμένου και δικηγόρου, ούτε η μεταξύ του επικοινωνία περιορίζονται κατά τρόπο που να φύγει τα δικαιώματα, την άσκηση των δικαιωμάτων τη υπεράσπιση. Προστασία απορρίτου. Υπογραμμίζουμε ότι υπάρχει το απόλυτο απόρριτο το, στις σχέσεις και για κάθε μορφή επικοινωνίας του δικηγόρου με τον ύποπτο ή με τον πελάτη του Επίσης 17, 19 και 27 τροπολογίες σε σχέση με τις ε, προξενικές αρχές. Λέμε ότι δεν θα πρέπει αυτές να χαίρουν ειδική μεταχείρισης ή παρεκκλήσεων, διότι δεν προβλέπεται στη σχετική σύμβαση της Βιέννης τέτοιου είδους παρέκκληση. Οποιαδήποτε παρέκκληση τους ή άλλους θα πρέπει να είναι περιορισμένη σε μόνο εξαιρετικές περιστάσεις. και η σχετική διευκρίνηση, η επαλήθευση θα πρέπει να γίνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση. Αν υπάρχει δηλαδή λόγος για παρέκκληση. Σε περίπτωση Φερρυπίν απαγωγής. Εάν και εφόσον ε, συμφωνούμε ότι είναι κατεπίγοντα τα μέτρα αυτά και με βάση τροπολογίες που έχουμε καταθέσει, θα πρέπει η απόφαση που θα, που θα μάλλον θα ανέβαλε το δικαίωμα για πρόσβαση σε δικηγόρο ε, να λαμβάνεται από δικαστικές αρχές. Και εφόσον προβλέπονται κατάλληλα ένδικα μέσα. Σε περίπτωση κινδύνου συνενοχής συνέργειας μεταξύ δικηγόρου και υπόπτου και πάλι θεωρώ ότι δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο να στερηθεί ο ύποπτο το δικαίωμα σε ε, υπηράσπιση σε δικηγόρο. Απλώ θα ήταν σκόπιμο να αντικατασταθεί ο ύποπτο για συνέργεια δικηγόρο με κάποιον άλλον. Στην παρουσία του δικηγόρου θεωρώ ότι είναι υπερβολική απέτηση να είναι παρόν δικηγόρος ακόμη και όταν ο ύποπτο ή κατηγορούμενο παρετείται του δικαιώματο αυτού. Πάντως πρέπει να ενημερώνεται ο ύποπτο ή κατηγορούμενο, του ε, τι συνεπάγεται η παρέτηση από το δικαίωμα στην υπεράσπιση από δικηγόρο. Αλλά επαναλαμβάνω, θα ήταν υπερβολικό να επιμείνουμε να υπάρχει δικηγόρο ακόμη και όταν παρετείται ο ύποπτο ή κατηγορούμενο. Τώρα για την ε, νομική αρρωγή, δηλαδή δωρεάν προσφορά δικηγορικών υπηρεσιών παρε... τη διαγράφουμε την πρόταση αυτή από το κείμενο με την τροπολογία 23 στο άρθρο 12 διότι θεωρούμε ότι θα επέβαλε ε, υπερβολικούς περιορισμούς στη δράση των κρατών μελών. Ίσως μπορούμε να το ξανασυζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί θα μπορούσε να βρεθεί μια λύση σε μελλοντικό νομοθέτημα το οποίο όμως θα αναφερόταν στη δικαστική αρρωγή συγκεκριμένα. Και θα καταθέσω τη σχετική τροπολογία. για την δωρεάν δικαστική αρρωγή. Για τον ορισμό του όρου του δικηγόρου έχω καταθέσει τροπολογία επίσης, καθώς γίνεται λόγος για το δικαίωμα σε δικηγόρο. Λέμε ότι αυτό είναι με βάση τον ορισμό των κρατών μελών για τη δικαστική αρρωγή σε συνήγορο. Αντίστοιχα η Επιτροπή των Νομικών Υποθέσεων έχει προτείνει έναν ορισμό για το, τι για το για το δικηγόρο, για την έννοια του δικηγόρου και πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε μια κύριη λύση. Αυτά είναι τα κύρια σημεία της εκθεσής μου και ευχαριστώ πολύ την Επιτροπή και το Συμβούλιο με τις δύο του προεδρίες οι οποίες κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες προκειμένου να προωθήσουν την υπόθεση αυτή και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις εισηγητές για τη συνεργασία. Ιδιαίτερα ευχαριστώ την Ιδανική Προεδρία για το ερωτηματολόγιο, την πρωτοβουλία να αποστείλει ένα ερωτηματολόγιο προ αρχή των κρατών μελών προκειμένου να διευκρινίσει τα διάφορα στοιχεία αυτή τη οδηγία, γιατί μα βοήθησε πολύ με τι πληροφορίε που συνέλεξε. Για το χρονοδιάγραμμα. Οι συνάδελφοι έχουν συμφωνήσει να παραταθεί η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών. Θα δω μαζί, σε συνεργασία με τη Γραμματεία ε, τι δυνατότητε υπάρχουν. Ευχαριστώ πολύ και περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστώ κύριε Αντωνέσκου για την παρουσίαση σας. Είναι σημαντικό το θέμα για τα δικονομικά δικαιώματα του υπόπτου ή κατηγορουμένου. Περιμένουμε να ακούσουμε τώρα τους συναδέλφους που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη συζήτηση. Πρώτα όμως νομίζω ότι θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, η Επιτροπή όχι, αλλά το Συμβούλιο ίσως να δουκουσουμε τωρα τους συναδελφους που ενδιαφερονται να κάνει κάποια σχόλια, εάν μου επιτρέπετε. Να δώσω το λόγο σύντομα στο Συμβούλιο Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την κυρία Αντωνέσκου. Με μεγάλη χαρά ε, έρχομαι εδώ να, σας, να εκπροσωπήσω το Συμβούλιο Ενώπιών σας για την ε, συζήτηση αυτού του σχεδίου εκθέσεως. Με μεγάλη χαρά επίσης ακούμε εκ μέρους της Προεδρίας ότι το ερωτηματολόγιο που ε, φτιάξαμε φάνηκε χρήσιμο στο Κοινοβούλιο. το Συμβούλιο με ικανοποίηση διαπιστώνει ότι η έκθεση εν γέννη έχει πορεία αντίστοιχη με αυτή των προπαρασκευαστικών εργασιών στο επίπεδο Συμβουλίου, πράγμα το οποίο θα μα βοηθήσει στη συνεργασία μα. Βλέπουμε δηλαδή με χαρά ότι το Συμβούλιο, όπω και η συγγήτρια, θεωρούν ότι η δυνατότητα για το δικηγόρο να επαληθεύει τι ε, συνθήκε κράτηση πρέπει να διαγραφεί από το σχέδιο προτάσεω δεδομένου ότι ξεπερνά το ε, πεδίο εφαρμογής και το στόχο του σχεδίου οδηγίας. Επίσης θα γνωρίζετε ότι οι διαπραγματεύσει στο Συμβούλιο για το σχέδιο οδηγίας δεν ήταν απρόσκοπτες. Έχουμε προχωρήσει τώρα και προχωρούμε καλά, αλλά υπάρχουν κάποια ζητήματα που δεν έχουν επιληθεί ακόμα και για το οποίο θα πρέπει να εξευρεθεί λύση. Μία από τις κύριες προκλήσεις είναι ότι τα τωρινά συστήματα για το δικαίωμα προσβάσης σε δικηγόρο στα κράτη-μέλη έχουν πολύ σημαντικές διαφορές από το ένα κράτος στο άλλο και ως εκ τούτου δεν θα είναι εύκολο να βρεθεί λύση αποδεκτή στους πάντες. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα, μια ιδέα δηλαδή ζητημάτων που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Στα παραπτώματα υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία θεωρούν ότι για τα μέτρα κατηγορίας Α και Β ε, πρέπει να έχουμε τον αποκλεισμό και στην τωρινή οδηγία, ο οποίος αποκλεισμός όμως δεν λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι για ορισμένα ακόμα και τροχαία παραπτώματα, όπως ε, ε, στάθμευση αυτοκινήτου σε χώρο που δεν επιτρέπεται η στάθμευση, ανήκουν στην αρμοδιότητα των ποινικών αρχών. Και ως εκ τούτου η διαδικασία πριν από τη δίκη, προανάκριση, ανάκριση από τις αρμόδιες αρχές, πάλι θα πρέπει να αποκλείεται. Αυτό λένε κάποια άλλα κράτη-μέλη. Κάποια άλλα κράτη-μέλη επίσης ως προς το περιεχόμενο και τη φύση της πρόσβασης σε δικηγόρο διαφοροποιούνται. Δηλαδή τι σημαίνει πρόσβαση σε δικηγόρο. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις σε κάθε περίπτωση ή μήπω θα πρέπει για ορισμένες περιπτώσεις να προβλέπονται πιο αυστηρές υποχρεώσεις. Φερρυπίν στην περίπτωση όπου κατηγορούμενος ή υποπτός μπορεί να του ή μπορεί να εμπλέκεται σε διαδικασίες ε, πριν από την παραπομπή του στο δικαστήριο. Ε, εν πάση περιπτώσει, θα είναι πολύ δύσκολο το έργο τη εξέφραση τη λεπτή ισορροπία που θα ικανοποιεί όλα τα κράτη-μέλη. Λεπτή ισορροπία η οποία θα πρέπει και τα δικαιώματα του υπόπτου και κατηγορουμένου να διαφυλάσει και να εξασφαλίζει όμως ταυτόχρονα τη δυνατότητα για τις αρχές δίωξης, τις δικαστικές αρχές να επιτελέσουν το έργο τους κατά τρόπο αποτελεσματικό που στη τελευταία ανάλυση πάλι σημαίνει προστασία των δικαιωμάτων του θύματος ενός εγκλήματος, μιας εγκληματικής πράξης. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε μια κοινή λύση μεταξύ των κρατών μερών επί τη βάση της προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πριν από το τέλος Προεδρίας μας εφόσον ε, εξασφαλιστεί με τη συμφωνία, θα μπορέσει να αποτελέσει βάση ε, συνεργασία διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που ξέρω δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Ωστόσο, η Προεδρία είναι βεβαία ότι θα διεξαχθεί η ε, διαπραγμάτευση αυτή σε πολύ καλές συνθήκες και προς όφελος όλων των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ θερμά για την προσοχή σα. Η Επιτροπή τελικά θέλει να σχολιάσει. Παρακαλώ, σύντομα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα την εισηγήτρια την κυρία Αντωνέσκου για την πρόταση αυτή. Έχουμε αναλύσει το σχέδιο έκθεσης, όπως επίση και τη Ζούρη, και όλα αυτά δείχνουν ότι η Επιτροπή πολύ σωστά στην πρότασή της περιλαμβάνει υψηλέ προδιαγραφές ασφάλεια για τα άτομα τα οποία κατηγορούνται, διώκονται. Βασιζόμαστε τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διατηρήσει ένα καλό επίπεδο δικαιωμάτων στην ε, οδηγία, υψηλό επίπεδο, ιδιαίτερα όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή, όπως είπε και η κυρία Αντωνέσκου, που ε, πρέπει να βοηθάει όλα τα άτομα, είτε αυτά κρατούνται είτε δεν κρατούνται, από τη στιγμή που κατηγορούνται για κάτι. Το περιεχόμενο που αναφέρεται στο δικηγόρο πρέπει να είναι πραγματικό, να μπορεί πραγματικά να υπερασπιστεί τον ε, πελάτη του και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στις εξαιρέσεις που πρέπει να είναι περιορισμένες και τις κυρώσεις από την άλλη μεριά σε περίπτωση που έχουμε παραβιάσεις ε, των όσων περιλαμβάνονται στην οδηγία. Αν υπάρχουν ε, πολλές ε, εξαιρέσεις και λίγες προβλέψεις δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Εμείς πάντως συμμεριζόμαστε τη φιλοδοξία να καταλήξουμε γρήγορα οι συνομοθέτες δηλαδή, σε συμφωνία και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε εμείς από την πλευρά μας για να διευκολύνουμε μια τέτοια συμφωνία. Ευχαριστώ. Ωραία. Συζήτηση τώρα. Πρώτος, η κυρία Ρομέρο Λόπες είναι η πρώτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ειλικρινά, πρόκειται για μια σημαντική πρόταση οδηγίας, γιατί μέσα στο πακέτο των δικονομικών δικαιωμάτων πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές οδηγίες. Η... Είναι τελευταία εξάλλου που έχει να κάνει με τα δικονομικά δικαιώματα που ξεκίνησαν με την Σουηδική Προεδρία. Χαιρόμαστε που έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει και ελπίζω να εγκριθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για μία πρόταση οδηγίας δύσκολη. Γιατί όπως είπε και ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, η κατάσταση από χώρα σε χώρα διαφέρει. Ο καθορισμός λοιπόν κάποιων ελάχιστων προδιαγραφών καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δύσκολο εγχείρημα. Πρέπει όμως παρόλα αυτά να τα καταφέρουμε και το δικαίωμα του κατηγορούμενου να είναι ένα πραγματικό και να εφαρμόσετε σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπει η οδηγία για να μην πω και σε περισσότερες ακόμα. Η κυρία Ντονέσκου έχει κάνει εξαίρετη δουλειά. Λίγα πράγματα θα μπορούσε κανείς να προσθέσει ενδιαφέροντα στις δικές της τις τροπολογίες. Πάντως επιμένουμε στη γραμμή που λέει ότι πρέπει να ενισχυθεί το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο και αυτό να γίνεται όσο γίνεται πιο γρήγορα στη διαδικασία. Από τη στιγμή δηλαδή που κατηγορείται κάποιος και πριν από τις ανακρίσεις. Όσον αφορά τώρα το δικαίωμα επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της κράτησης, είναι προφανές ότι και εδώ πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ο ύποπτος ευθύς εξ αρχής να μπορεί να δέχεται επισκέψεις από, τους, από την οικογένειά του, τους συγγενείς του. Όσον αφορά τώρα το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο, πιστεύουμε ότι εδώ είναι σημαντικό η παρουσία του δικηγόρου να διασφαλίζεται να υπάρχει εγγύηση για αυτήν δηλαδή. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει δυσκολία με τα αποδεικτικά στοιχεία. Ο δικηγόρος δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει πάντα ως εγγύηση. Το θέμα του απορρίτου τώρα της εμπιστευτικότητας είναι επίσης κάτι που πρέπει να στηρίξουμε. Στην Ισπανία, τελευταία, είχαμε αποφάσεις δικαστικές, οι οποίες έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτό το σημείο. Πώς δηλαδή υποστηρίζουμε τα δικαιώματα του κατηγορούμενου. Προσοχή πότε θα υπάρχει εξαίρεση στην εμπιστευτικότητα. Γιατί η παραβίαση του απορρίτου στη σχέση δικηγόρου και πελάτη του, καταλαβαίνετε, πρέπει να ισχύει μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις, σε πραγματικές εξαιρέσεις και πρέπει να δούμε ποιες θα είναι αυτές οι έκτακτες περιπτώσεις οι οποίες θα επιτρέπουν την παραβίαση αυτού του δικαιώματος στην εμπιστευτικότητα. Συνέβη στην Ισπανία και σίγουρα και σε άλλες χώρες, είναι πιθανόν οι δικηγόροι τελικά να ασκούν το καθήκον του της υπεράσπισης, αλλά με κάποια συνενοχή με τον πελάτη του. Τότε όμω δεν πρόκειται για δικηγόρο, τότε πρόκειται για κάτι άλλο. Αν υπάρχει απόδειξη ότι οι δικηγόροι μπορεί να μην κάνουν τη δουλειά τους, αλλά να κάνουν άλλη δουλειά, τότε εννοείται ότι πέρα από το θέμα του απορρίπτου υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει. Θέλω να πω ότι είναι δύσκολο να καθοριστούν οι εξαιρέσει. Θα προσπαθήσουμε πάντως. Όσον αφορά το άρθρο 8 που μιλάει για τις εξαιρέσει, το δικαίωμα υπεράσπισης έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να πληγεί με τίποτα. Για το άρθρο 12 τώρα όσον αφορά τη δικαστική αρρωγή δωρεάν. Εδώ δεν ξέρω αν θα βγει από τις δικονομικές εγγύσεις γιατί υπάρχουν ελάχιστες προδιαγραφές πρόσβασης οικονομικές για παράδειγμα. Γιατί ορισμένοι πιθανόν να μην μπορούν να πληρώσουν έναν δικηγόρο. Το δικαίωμα αυτό δηλαδή δεν είναι δικαίωμα αν δεν λαμβάνει υπόψη και αυτή την πτυχή της αδυναμίας πληρωμής. Γι' αυτό πρέπει να διασφαλιστεί η ελάχιστη δικαιοσύνη σε κάθε χώρα για την ε, δωρεάν πρόσβαση σε δικηγόρο. Φυσικά και οι περιπτώσεις διαφέρουν από χώρα σε χώρα, οπότε και αυτή τη δωρεάν πρόσβαση σε δικηγόρο πρέπει πολύ προσεκτικά να δούμε τι τροπολογίες μπορούμε να υποβάλουμε εδώ. Ξέρω ότι το σκέφτεται και η συγγήτρια, κυρία Αντωνέσκου. Πρέπει να προχωρήσουμε ακόμα πιο πολύ πάντως σε σχέση με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που λέει να ξεχωριστεί το θέμα αυτό από τις δικονομικές εγγύσεις. Ευχαριστώ. Περνάμε στην κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι η κυρία Αντωνέσκου, όπως ήταν αναμενόμενο, έκανε μια πολύ καλή δουλειά και μας παρουσίασε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα με το οποίο εν πολύ συμφωνώ. Το βασικό άρθρο είναι το 3 και νομίζω ότι έχει δίκιο που βασίζεται στο δικαίωμα παρουσίας δικηγόρου κατά τη διάρκεια της ανάκρισης από πλευράς των αστυνομικών αρχών. Για το εάν τώρα η λέξη interview στα αγγλικά είναι η σωστή λέξη, δεν ξέρω αν σημαίνει εθελοντική παρουσία προσώπου στο αστυνομικό τμήμα ή κάτι άλλο, αυτό πρέπει να διευκρινιστεί. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι όταν κάποιος καθίσταται ύποπτος ή χαρακτηρίζεται ύποπτος ή χαρακτηρίζεται ακόμα περισσότερο κατηγορούμενος, το θέμα είναι αν σε αυτή την περίπτωση δεν ισχύει η προηγούμενη ρύθμιση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έλεγα απαιτεί περισσότερη εξέταση. Το βασικό θέμα σε αυτή την οδηγία, το οποίο δεν έχει ακόμα επιληθεί διότι έχει δυσκολίες στο Συμβούλιο, είναι ότι όχι μόνο υπάρχει το δικαίωμα του υπόπτου να ζητήσει την παρουσία δικηγόρου, αλλά υπάρχει υποχρέωση του κράτους να καταστήσει διαθέσιμη την παρουσία δικηγόρου, να διαθέσει δικηγόρο και αν δεν διευκρινιστεί και δεν επιληθεί αν θέλετε αυτό το συγκεκριμένο θέμα τότε κινδυνεύουμε να καταλήξουμε με μια οδηγία η οποία στα χαρτιά θα είναι καλή αλλά πρακτικά δεν θα λειτουργεί. Το πρόβλημα λοιπόν το οποίο θα πρέπει να λύσουμε είναι ότι πολλές χώρες μέλη πληρούν την περιπτωσιολογία αν θέλετε και την ομολογία του ε, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Από την άλλη υπάρχουν περιπτώσεις όπου έχουν γίνει ανακρίσεις και εξετάσεις υπόπτων χωρίς την παρουσία δικηγόρου. στο νομικό σύστημα της χώρας από την οποία προέρχομαι, το πρόβλημα αυτό έχει οδηγήσει σε υποτιθέμενες ομολογίες και έχουν υπάρξει επί τη βάση αυτών των υποτιθεμένων ομολογιών αποφάσεις οι οποίες ήταν εντελώς λανθασμένες από πλευράς των δικαστηρίων. Λοιπόν, το θέμα της εξέτασης ή της ανάκρισης ενός κρατουμένου ή ενός υπόπτου είναι κάτι το οποίο πρέπει να πλαισιωθεί με συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι αλλαγές προτείνει ή θα προτείνει η κυρία Αντωνέσκου σε σχέση με τις προτάσεις του Συμβουλίου. Πάντως θα συμφωνήσω με την κυρία Αντωνέσκου ότι το συγκεκριμένο αυτό μέτρο ε, δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των θεμάτων που αφορούν τη νομική αρρωγή, αλλά ή την νομική συνδρομή καλύτερα. Αλλά το γεγονός είναι ότι τίθεται ένα ερώτημα. Έχει υποχρέωση το κράτος μέλος να παράσχει δικηγόρο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες. Αν δεν διευκρινιστεί αυτό, τότε μόνο οι πλούσιοι σαν παράδειγμα σε κάποιες περιπτώσεις θα έχουν ε, νομική βοήθεια και δεν θα υπάρχει βοήθεια του κράτους ε, για την παρουσία δικηγόρου. Ή από την άλλη αν επιτρέπεται η παρουσία δικηγόρου αλλά δεν, δεν διευκρινίζεται ότι το κράτος έχει την υποχρέωση να συνδράμει στην έβρεση του δικηγόρου αυτό πάλι είναι θα έλεγα κάτι το οποίο αναιρεί στην ουσία την πρόταση. Η κυρία Αντωνέσκου έχει επιδείξει την απαιτούμενη ευελιξία λοιπόν σε σχέση με την παρουσία δικηγόρου σε σχέση με τη συλλογή αποδείξεων ή τεκμηρίων. Νομίζω ότι το αρχικό, το αρχικό κείμενο της Επιτροπής δεν προσέφερε ε, πολλά σαν παράδειγμα στην παρουσία δικηγόρου όταν η αστυνομία ε, προχωρούσε στη συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων. Αλλά υπάρχουν άλλες ε, καταστάσεις στις οποίες άλλες δραστηριότητες ανακριτικές της αστυνομίας και συλλογή τεκμηρίων όπου η παρουσία δικηγόρου θα μπορούσε να είναι χρήσιμη. Και γι' αυτό νομίζω ότι η πρόταση Αντωνέσκου είναι καλή. Θα συμφωνήσω επίσης και με το Συμβούλιο και την κυρία Αντωνέσκου σε σχέση με τον ρόλο των δικηγόρων <clears throat> στην κρίση και την αξιολόγηση των συνθήκων κράτησης. Εκεί δεν έχει σημασία ο ρόλος του δικηγόρου. Θα έλεγα υπάρχουν άλλες αρμόδιες υπηρεσίες σχετικά με την εμπιστευτικότητα Κυρία Λάτφορντ, πρέπει να επιταχύνουμε λίγο γιατί 12.30 πρέπει να τελειώσουμε και έχουμε ακόμα πολλούς που θέλουν να μιλήσουν. Λέγεται εδώ ότι η εμπιστευτικότητα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκλείει την δυνατότητα να υπάρχουν ε, ε, σωματικές έρευνες, σαν παράδειγμα, χωρίς παρουσία δικηγόρου. Εδώ θα πρέπει να είμαι λιγότερο απόλυτη από την κυρία Αντωνέσκου και θα συμφωνήσω ε, με τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου που λέγει ότι θα πρέπει να υπάρχει σωστός χρονισμός Έχει επίσης δίκιο στην τροπολογία 8 η κυρία Αντωνέσκου, όπου ζητάει για πιστοποιημένους ε, εκπροσώπους δικηγορικών γραφείων, οι οποίοι δεν είναι δικηγόροι αλλά είναι εκπαιδευμένοι έτσι ώστε να δίδουν νομικές συμβουλές. Και επίσης να προβλέψουμε και τις συνθήκες σχετικά με την παροχή ε, συνδρομής μέσω τηλεφωνικής συνδιάλεξης. Λοιπόν, δεν θα κάνω κάποιο άλλο σχόλιο. Νομίζω ότι η κυρία Αντωνέσκου μας έδωσε μια σωστή πλατφόρμα, αν θέλετε, πίτευξη συμφωνίας με το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο όμως θα πρέπει να δώσει μια κάποια λύση ε, στο τι σημαίνει στην πρακτική η παρουσία του δικηγόρου και ποιος πραγματικά είναι ο ρόλος που διασφαλίζει την παρουσία του δικηγόρου. Κοιτάξτε, έχουμε άλλους δύο σκιώδεις εισηγητές και κάποια μέλη. Λοιπόν, παρακαλώ, ε, κοιτάτε, 12 και μισή, έτσι και αλλιώς 12.30 θα τελειώσουμε για σήμερα το πρωί. Ο κύριος Ντε έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ πολύ τον, ε, την εισηγήτρια. Πιστεύω ότι είναι μια καλή βάση για να ξεκινήσουμε. Εγώ θα επιμείνω για την ισορροπία. Από τη μια στιγμή υπεράσπιση που χρειάζεται και από την άλλη μεριά ε, να προχωρήσει η διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν και με απασχολεί πολύ το θέμα των μικρών ε, προβλημάτων των μικρών ε, εγκλημάτων. Και θέλω τόσο συζητάμε εδώ να ξεκινάνε από την πρώτη στιγμή. Ε, δηλαδή πριν καν απαγγελθεί κατηγορία. Εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει δικηγόρος. Η κυρία Τονέσκου το προσπαθεί αυτό. Τώρα για το θέμα του απορρίτου. Συμφωνώ με την εισηγήτρια για το ότι βασικό είναι όπως λέει και η κυρία Λάτφορτ υπάρχουν περιπτώσεις που μερικές φορές ε, ο δικηγόρος δεν κάνει τη δουλειά του. Για το ρόλο λοιπόν του δικηγόρου εδώ Δυστυχώς έχουμε διάφορες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν και με το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, όπου τα πράγματα δεν πήγαν καλά και όπου ήταν προβληματική η κατάσταση για τον κατηγορούμενο. Πιστεύω λοιπόν ότι γι' αυτό πρέπει να υπάρχει ο δικηγόρος, γιατί έχει ένα πραγματικό ρόλο. Τέλος, συμφωνώ με το ότι είναι ένα μέσο που έχουμε στη διαθεσή μας, ώστε όντως να υπάρχει το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο, είναι μια καλή ρύθμιση, αλλά χρειαζόμαστε και κάτι άλλο που είναι η υπεράσπιση του κατηγορούμενου. Ίσως να χρειάστηκε κάτι άλλο και καλό θα ήταν να το συμπεριλάβουμε αυτό στο προήμιο. Ελπίζω όσο γίνεται πιο γρήγορα ε, σχετικά με την δικαστική αρρωγή θα έχουμε πρόοδο. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ για άλλη μια φορά ευχαριστώ την εισηγήτρια, την καλή συνεργασία μέχρι τώρα. Ήθελα να επισημάνω δύο σημεία που θεωρούμε σημαντικά πάντα. παρουσία συνηγόρου κατά τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. όπου θα θέλαμε να είναι πιο σαφή η διατύπωση, όπως και στη δυνατότητα για τον δικηγόρο να επαληθεύσει τις συνθήκες κράτησης, εφόσον έχει επιβληθεί η στέρηση ελευθερίας του αυτό λοιπόν θα θέλαμε να διευκρινιστεί, να εξασφαλιστεί η πρόσβαση του δικηγόρου, η επαλήθευση και επίση την τροπολογία υπαριθμών 21 που έχουμε καταθέσει. Και στην οποία επιμένουμε, διότι πρόκειται για την συνεργασία και σε περιπτώσεις ε, παρουσίας του δικηγόρου, όταν έχουμε να κάνουμε διεθνές ένταλμα ή έρευνα ή κράτηση. Και εκεί θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης του ε, δικηγόρου. Ευχαριστώ κύριο Και πρέπει να πω ότι δεν χρεώνω το λεπτό σήμερα, μιλάω όσο θέλω δηλαδή. Ε, θα ήθελα να υποστηρίξω τις ε, γενικότερες αρχές, τις γενικές αρχές, μπορούμε να τις δεχθούμε. Υπάρχουν προτάσεις ικανοποιητικές, Απλώς, ως προς παρατηρήσεις κυρίας Λάτφορτ για την ε, θέση του δικηγόρου ή του παραδικηγορικού προσωπικού, paralegal, ε, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς τη χρήση αυτής της ορολογίας, διότι paralegal είναι μια έννοια πολύ διαφορετική σε κάθε κράτος μέλος. Πρόσβαση λοιπόν στο δικηγόρο, ναι βεβαίω, αλλά πρόσβαση σε κάποιον ο οποίο έχει μερικέ μόνο ή και καθόλου γνώσει γνώσεις ε, νομικές και απλώς εξυπηρετεί ως βοηθός έναν δικηγόρο πρέπει να είναι μια διαφορετική υπόθεση. Για το κόστος τώρα, το κόστος, η δαπάνη, δεν θα πρέπει να επιβαρύνει πάντοτε το κράτος για την πρόσβαση στο δικηγόρο πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να το δούμε το θέμα αυτό και πολύ μεγάλη ευαισθησία. Ιδάλλως δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με σαφήνεια όπως το θέλαμε. Αλλιώς τίποτα άλλο δεν έχω να προσθέσω. Ευχαριστώ και συγχαίρω ιδιαίτερα την εισηγήτρια για τη δουλειά της. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ήσταν ιδιαίτερα σύντομο. Για να δούμε τώρα τους λοιπούς συναδέλφου που ενδεχομένω θέλουν να λάβουν το λόγο. Κύριε Μπουζούτη, εσείς πρώτο. Πρόεδρε, ευχαριστώ και ξεκινώ ε, συγχαίροντας την κυρία Αντωνέσκου όπως και συναδελφή εξαιρετική δουλειά και πολύ προσεκτική και ισορροπημένη η προσέγγιση της. Αυτό το βλέπουμε και συγκεκριμένα στην εφαρμογή στην ε, χώρα μου που διαφοροποιείται από άλλες, όπως υποδείχθηκε και νωρίτερα. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να ε, προχωρήσουμε με βάση αυτές τις προτάσεις. Μπορούν να αποτελέσουν δηλαδή μία βάση, μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Ε, θέση εφαρμογή των σαφέστατων όσον αφορά την πρόσβαση, το δικαίωμα για πρόσβαση σε δικηγόρο, ε, αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ε, επίσης κάποια άλλα σημεία που επεσήμεναν ε, συνάδελφοι που θα ήθελα να υπογραμμίσω πολύ σύντομα ε, στις λιγότερο σημαντικές υποθέσεις ή στη συζήτηση για το ποιες είναι οι υποθέσεις που θα πρέπει να αποκλείονται. Είναι σημαντικό νομίζω να μην υποβιβάζουμε τα θέματα αυτά λέγοντας ότι πρόκειται για λιγότερο σημαντικές υποθέσεις ε, και θα πρέπει να μείνουν εκτός πεδίου εφαρμογής. Επίσης, σε ποιο σημείο της διαδικασίας αρχίζει να εφαρμόζεται, να ισχύει το δικαίωμα για προσβάση δικηγόρο. Αυτό που θα εξαρτηθεί από το ποιο είναι το χρονικό σημείο από το οποίο κανείς θεωρείται κατηγορούμε, ύποπτο μάλλον, δηλαδή πότε αρχίζουν, γιατί νομίζω ότι είναι ξεκάρα, ξεκάθαρο ότι άπαξ και επαγγελθούν κατηγορίε, πρέπει να οπωσδήποτε να εφαρμόζεται το δικαίωμα, να το δικαίωμα τη πρόσβαση. Μετά, σε περίπτωση καθυστερήσεων ή περιορισμού των ερευνητικών διαδικασιών και δισεπινικές ε, περιπτώσεις. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να βρούμε τη χρυσή τομή. Και τέταρτον, νομική αρρωγή, δωρεάν δικηγορική αρρωγή. Θα συμφωνήσω περισσότερο με την κυρία Αντωνέσκου ότι μια και η νομική αρρωγή έχει τέτοιο λεπτό και σημαντικό χαρακτήρα, θα έπρεπε να παρακαλέσουμε την Επιτροπή, πιστεύω, να αφήσει το θέμα αυτό για μια χωριστή αντιμετώπιση, έτσι ώστε να μην χαθεί μέσα στη γενικότερη συζήτηση της τρέχουσας οδηγίας. Είναι πολύ σημαντικό φυσικά όταν προβλέπετε δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο να είμαστε και βέβαιοι ότι θα εφαρμόζεται πράγματι σε όλους το δικαίωμα αυτό και ιδιαίτερα σε αυτούς που το έχουν προς ανάγκη. Όμως και με δεδομένο ότι προβλέπεται μια σχετική πρόταση, ας αφήσουμε να ρυθμιστεί η ε, δικαστική αρρωγή σε, την, ε, σε αυτό το πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Φως. Πρόεδρε, στην ε, στο δικαίωμα για πρόσβαση σε δικηγόρο, η δικαστική αρρωγή αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Εξασφαλίζει την ουσιαστική προσφορά δικηγορικών υπηρεσιών περάσπισης. Είναι πολύ καλή έκθεση της κυρία Αντωνέσκου, πολύ καλά εξισορροπημένη, ιδιαίτερο ο τομέας, το πεδίο εφαρμογή τη οδηγία που έχει προσδιορίσει και ο αποκλεισμό τη δωρεάν δικαστική αρρωγή μου φαίνονται πολύ θετικά στοιχεία. Κάποια σημεία που θα ήθελα να προτείνω για συζήτηση συνθήκες κράτησης, απόρριτο και απαγόρευση ε, υποβάθμισης. Θα ήθελα να συζητήσω με την εισηγήτρια, όπως άλλωστε το έχω κάνει και νωρίτερα, στα άρθρα 12 και 13, 2, την δυνατότητα που προβλέπεται να επαφηθεί το θέμα αυτό στα κράτη-μέλη. Στο απόρριτο, τροπολογία 36, βεβαίως εν γέννη οι διαβουλεύσεις μεταξύ δικηγόρου και πελάτη ε, κατηγορουμένου είναι δεδομένες. Αλλά υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου μπορεί να επιτρέπεται η παραβίαση του απορρίτου όταν υπάρχουν σοφαρές εικόνες, σε παραδείγματι ότι μπορεί να υπάρχει εγκληματική ε, συνέργεια μεταξύ πελάτη και δικηγόρου ή αν ε, μπορεί να ε, κινδυνεύει η ζωή ή η ελευθερία κάποιου τρίτου προσώπου. Έτσι λοιπόν έχουμε τις τροπολογίες 41 όπου το δικαίωμα του κατηγορουμένου για την επαλήθευση των συνθήκων κράτησης προβλέπεται από την πρώτη Ευρωπαϊκής Επιτροπή, αλλά η συγγήτρια προσπαθεί να ενισχύσει το περιεχόμενο του δικαιώματος πράσβεσης, δεν βλέπω κανένα πρόβλημα σε αυτό, για δε το Συμβούλιο, για τα παραπτώματα είναι μία έννοια η οποία ε, έχει βρει την ε, θέση της μέσα στις ε, διαδικασίες ώστε να μην θεωρείται ποινικό αδίκημα κάθε ελάχιστο παράπτωμα ή πτέσμα και νομίζω ότι είναι καλό να αποκλειστούν από αυτές τις υποθέσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σπίρκερ, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Αντωνέσκου και να εκφράσω την υποστήριξή μου προς τις προτάσεις της με δύο-τρεις μόνο παρατηρήσεις και προτάσεις για τροποποίηση στην 28 τροπολογία του άρθρου, για το άρθρο 3 συγκεκριμένα, το δικαίωμα της άμεσης ή ταχείας πρόσβασης σε δικηγόρο. Στο κείμενο της Επιτροπής λέγεται πριν από την ανάκριση, από την αστυνομία και άλλες αρχές, μήπως θα έπρεπε η πρόσβαση δικηγόρου να εξασφαλίζεται καλύτερα από την ανακριση απο την αστυνομια και αλλες αρχες μηπως θα επρεπε η προσβαση δικηγορο να εξασφαλίσετε καλυτερα απο την εναρξη της ανάκρισης, ώστε να είναι δυνατόν να λαμβάνεται η αυθεντική τοποθέτηση ε, του υπόπτου ή κατηγορουμένου και όχι εκείνη η οποία θα έχει διαμορφωθεί από τις συμβουλές ενδεχομένως του δικηγόρου του. Αυτό θα διευκολύνει βέβαια και, τις, και προς όφελος των θεμάτων τις ερευνητικές και ανακριτικές διαδικασίες. Νομίζω λοιπόν ότι η υπεράσπιση, η πρόσβαση δικηγόρου θα πρέπει να ξεκινάει από την ανάκτηση και όχι πριν από αυτή. Επίσης, από το άρθρο 4 παράγραφο 2 προβλέπεται, 2 προβλέπεται ότι θα πρέπει ο δικηγόρος να παρίσταται στην ανάκριση και να υποβάλει ερωτήσεις. Ε, ωστόσο, χωρίς να παρεμποδίζει τη συλλογή ε, αποδεικτικών στοιχείων. Εγώ θα πρότεινα ο δικηγόρος να έχει το δικαίωμα να παρίσταται μετά την συλλογή αποδεικτικών, μάλλον μετά από τη συλλογή αποδεικτικών να διατυπώνει ερωτήσεις Πρώτα δηλαδή να γίνεται η συλλογή των στοιχείων. Στο απόρριτο, συμφωνώ με τον κύριο Φως, ότι ναι βεβαίως εν γέννη πρέπει να εξασφαλίζεται, αλλά όχι απόλυτα και για κάθε συνάντηση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη και πάντως όχι όταν υπάρχει προσπάθεια όταν διαγιγνώσκεται μια προσπάθεια απόκρυψης στοιχείων ή ε, παραχάραξη στοιχείων. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις δηλαδή θα μπορούσε να οδηγήσει ε, ο κίνδυνος να αλλοιωθούν τα αποδεικτικά στοιχεία και σε άρση του απορρίτου Τη της επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρου και ε, πελάτη του. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα, πέρασε ο χρόνος. Πριν περάσουμε πίσω στην κυρία Αντωνέσκου, παρακαλώ εσείς. Ευχαριστώ και εγώ την ε, συνάδελφο, λέει η κυρία Γρίσβεκ για το κείμενό της. Βέβαια, για να μην μείνει ένα ωραίο έγγραφο, μία δήλωση προθέσεων, αλλά να υπάρχουν και οι να πετύχει, καλό θα ήταν με τροπολογίες να υπάρξει βελτίωση. Και να έχουμε και χρόνο, εάν θέλουμε ένα πραγματικό, πραγματικά κοινό σύστημα, το οποίο να επιτρέπει στα διαφορετικά νομικά μας συστήματα να λειτουργούν αποτελεσματικά με υψηλό επίπεδο δικονομικής προστασίας. Επί ουσίας πρώτα απ' όλα. Σε ορισμένε χώρες οι ποινικέ ε, διώξεις είναι πολύ πιο ευρύ πεδίο από τις άλλες χώρες και ε, το κείμενο θα έπρεπε να πετύχει μια καλή ισορροπία. Αλλά να είναι και αποτελεσματικό, να μπορεί να εφαρμοστεί. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να βρούμε τα μέσα, να πετύχουμε την ισορροπία αυτή, χωρίς να βάζουμε όλες τις παραβάσεις μαζί. Να δούμε τη διαφορά που υπάρχει στο γαλλικό σύστημα, για παράδειγμα, ανάμεσα στην ε, ε, ακρόαση και από την άλλη μεριά την ε, προσωρινή κράτηση. Καλό είναι λοιπόν να τα δούμε αυτά για να είναι αποτελεσματική η ρυθμισή μας. Θα ήθελα να δουλέψουμε περισσότερο σε βάθος για παράδειγμα και να κάνουμε τη διάκριση ανάμεσα στις διώξεις σε περίπτωση ανακρίσεων που έχουν να κάνουν με την τρομοκρατία το μεγάλο έγκλημα. Γιατί εδώ ίσως να υπάρχει ένα παραπάνω στοιχείο που να απαιτεί ταχύτητα και ίσως θα έπρεπε να το συμπεριλάβουμε. Τέλος, για την ε, νομική συνδρομή, η τροπολογία 23 που αναφέρεται σε αυτήν, ίσως δεν επιτρέπει σε όλα τα πρόσωπα να υποφελούνται από το δικαίωμά του στην υπεράσπιση. Και σε αντίθεση με τόσα πιστεύω ο συνάδελφος Κίφοφ και ο οποίος ανησυχεί για τα κράτη, μα ο στόχος των κρατών είναι ακριβώς να υπάρχει ισότητα μεταξύ όλων. Αυτό θα πρέπει να είναι ο τελικός στόχος των κρατών, ισότητα μεταξύ όλων των πολιτών και να εξυπηρετούν τους πολίτες. Θα υποφεληθώ από τη διαδικασία τροπολογιών. Πρόεδρος, ωραία. Έπρεπε να σταματήσουμε τώρα, αλλά η κυρία Τονέσκου, μια που έγινε τόση συζήτηση, παρακαλώ να είσαστε σύντομοι κι εσύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Θα επαναλάβω αυτό που είπε η κυρία Λάτφορτ, ότι δηλαδή πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε προδιαγραφές οι οποίες καθορίζονται από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και δεν μπορεί τώρα να τα παραβλέπουμε. Δεν μπορεί να αποφασίσουμε μια οδηγία η οποία να έχει κατώτερε προδιαγραφέ από αυτέ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είχαμε την περίπτωση κατά τη Τουρκία, σύμφωνα με την οποία η πρόσβαση σε δικηγόρο πρέπει να υπάρχει από την αρχή των ανακρίσεων, από το πρώτο στάδιο. Έλαβα, δοσημείωσα μάλλον όλα όσα είπαν οι συνάδελφοι για τα ελαφρά παραπτώματα, <clears throat> για το απόρριτο. Θα τα λάβω υπόψη μου και θα προσπαθήσω να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Τώρα για την 13. Ε, εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όσο υπάρχει υποχρέωση πρόσβαση σε ένα δικαίωμα, πρέπει να υπάρχουν και κυρώσει αν δεν διατίθεται το δικαίωμα αυτό, δεν προσφέρεται. Η διάταξη που είχαμε στο σχέδιο πρότασης έρχεται σε αντίθεση με τις νομικές παραδόσεις ορισμένων χωρών, είπαν κάποιοι. Ε, πρέπει λοιπόν να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να τα συμβιβάσουμε όλα αυτά. Ζητήσαμε γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας και την περιμένουμε. Πρέπει να βρούμε τον καλύτερο δυνατόν τρόπο για να ρυθμιστούν οι περιπτώσεις εκείνες όπου ένα κράτος αρνήθηκε στον ύποπτο την παρουσία δικηγόρου. Γιατί αυτό το οποίο έχουμε τώρα με την πρόταση της Επιτροπής είναι ότι οι αποδείξεις ή οι ανακρίσεις που έχουν γίνει εφόσον δεν έχει ληφθεί υπόψη το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο γίνονται άκυρες, καταστώνται άκυρες. Τώρα στον κύριο Άλμπρεχτ που μίλησε για την παρουσία δικηγόρου κατά τη διάρκεια συλλογής αποδείξεων. Με... Πιστεύω και εγώ ότι η τροπολογία σχετική μπορεί να βελτιωθεί. Όσον αφορά τώρα τον ορισμό του δικηγόρου, θεώρησα αναγκαίο να υπάρξει ορισμός αυτός, γιατί στόχος της οδηγίας είναι το δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο. Και δεν είναι εύκολο να βρει κανείς τον καλύτερο ορισμό ο οποίος να καλύπτει όλα τα νομικά συστήματα όλων των χώρων μελών. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να βρούμε τον καλύτερο τρόπο για να ορίσουμε το ότι είναι δικηγόρος. Και άλλη μια φορά σας ευχαριστώ πολύ όλους και ελπίζω να κατάφερα να ε, καθισχάσω τις ανησυχίες σας και από εκεί και πέρα ευχαρίστω σε ό,τι διάλογο θέλετε προκειμένου να καταλήξουμε σε συμβιβασμό. Είμαι στη διάθεσή σας. Μπράβο, λέω πρόεδρο, σε ευχαριστώ που ήσασταν σύντομοι. Σα ευχαριστώ και εγώ πολύ για τη δουλειά σα για την οποία σα συνεχάρισαν οι περισσότεροι από αυτού που πήραν το λόγο. Τώρα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Τέλη Μαρτίου να έχουμε τη συνέχεια. Συντονιστές τώρα. Συνεπώς, τι προτείνω. Προτείνω μόνο οι συντονιστές και όσοι έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην ιδρύαση των συντονιστών να παραμείνουν στην αίθουσα για την επόμενη ώρα. Οι υπόλοιποι ελεύθεροι. Μπορείτε να συνεχίσετε αν θέλετε πάντως τρεις η ώρα να είσαστε πίσω εδώ γιατί θα συνεχίσουμε με τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Please, let's haste